Καλησπέρα σε όλους. Παρακαλώ να, να καθίσετε. Για να ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση. Με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα ακούσουμε μια παρουσίαση του θεματικού τμήματος Α Ευρώπη, το Παγκόσμιο Κέντρο της Άριστης Έρευνας. Και έχουμε προσκαλέσει για το σκοπό αυτό την κυρία Βέκλερς, ε, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λεύεν, στο τμήμα ε, στρατηγικής και κοινοτομίας. Μάλιστα είναι ε, μέλος του Μπρίκερ από το 2009. Είναι μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου και από το 2004 έως το 2008 ε, είχε άδεια και ήταν σύμβουλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης έχει υπηρετήσει στο Επιστημονικό Συμβούλιο ερση για τέσσερα χρόνια καθώς και στην ομάδα εμπειρογνωμόνων όπου συμβούλευε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα έρευνας. θα μας παρουσιάσει μια έρευνα για τις δυνατότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτελέσει κέντρο αριστείας στην έρευνα. Η έρευνα επίσης εξετάζει πώς μπορούν οι δημόσιοι πόροι Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλλουν σε αυτό. Οι συντονιστές μας ζήτησαν τη μελέτη αυτή ως προετοιμασία για τις εργασίες μας πάνω στο ορίζον Ευρώπη. Οι συστάσεις στηρίζουν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την καθηγήτρια Βέκελες να ε, μας ξεκινήσει την παρουσίασή της. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή, καταρχάς να εκπονήσω τη μελέτη, αλλά και πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα. Ε, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επανέλθετε στην ίδια την έκθεση, οπότε δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Ε, θα σας παρουσιάσω τα βασικά συμπεράσματα. Όπως ήδη υπόθηκε κατά την εισαγωγή, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να διαπιστώσουμε τι δυνατότητες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει παγκόσμιο κέντρο ε, αριστείας στην έρευνα. Εξετάζουμε δηλαδή το τοπίο όσον αφορά την ε, τεχνολογία, την έρευνα ε, και να δούμε ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και πώς έχει συμβάλει το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό. Και έχω και κάποιες συστάσεις να σας δώσω, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι καλή ιδέα να εκπονήσουμε τη μελέτη αυτή διότι γίνονται σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο, στην παγκόσμια σκηνή. Έχουμε την ε, άνοδο της Κίνας ε, που αποτελεί νέο πόλο ε, δίπλα στους παλιούς πόλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι αυτό απειλεί τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι Μερικοί θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ε, μηδενικού αθροίσματος, δηλαδή ότι αν η Κίνα ανέβει θα πέσουμε εμείς, αλλά μπορεί, μπορούμε να το δούμε αυτό και ως ευκαιρία, διότι έτσι αυξάνεται το παγκόσμιο δυναμικό ε, στην επιστήμη και την τεχνολογία. Έτσι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε ε, νέα ταλέντα και να εμβαθύνουμε την έρευνα και να βελτιωθούμε σε τομείς όπου ούτως ή άλλως έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Επίσης, ε, έχουμε το πρόγραμμα πλαίσιο με τη νέα προοπτική του Horizon Ευρώπη αποτελεί λοιπόν καλή ευκαιρία να εξετάσουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά ή να πετύχουμε τους στόχους μας καλύτερα. Πολύ ε, σύντομα αρχικά θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω για τις νέες τάσεις όσον αφορά το παγκόσμιο τοπίο. Αλλά τα περισσότερα δεδομένα ούτως ή άλλως μπορείτε να τα βρείτε στην ίδια την έκθεση. Σημαντικό όσον αφορά τις τάσεις ε, είναι η αύξηση της Κίνας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πόσο γρήγορα ανεβαίνει όσον αφορά την έρευνα, την καινοτομία. Σε όλες τις διαστάσεις βλέπουμε σημαντική πρόοδο και ιδιαίτερα στον τομέα της επιστήμης κινείται πάρα πολύ γρήγορα και προκαλεί την ε, κοντεύει να φτάσει τις Ηνωμένε Πολιτείε που βρίσκονται στην πρώτη θέση. Και αν κοιτάξουμε συγκεκριμένου τομεί όπω είναι η μηχανική, τα υλικά, την υπολογιστική, βλέπουμε ότι η άνοδος της Κίνα είναι ακόμη πιο γρήγορη από τη γενική τη τάση και όχι μόνο όσον αφορά την ποσότητα. βλέπουμε όμως και πολύ σημαντική ε, άνοδο όσον αφορά την ποιότητα. Πιο σημαντικό θέμα λοιπόν είναι σε τι βαθμό αυτή η άνοδος νέων πόλων μπορεί να ωφελήσει άλλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ωφεληθεί από αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να επωφεληθεί από αυτήν την πολυπολικότητα Πιστεύουμε ότι μπορεί να υποφεληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτον μέσω της διεθνού συνεργασία, δηλαδή η Ευρώπη πώς μπορεί να συνεργαστεί με άλλους σημαντικούς πόλους της επιστήμης και πώς μπορεί να δημιουργήσει ε, δική, δικό της χώρο αριστείας. Πρόκειται λοιπόν για ένα εργαλείο για την αριστεία στην έρευνα. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η διεθνής κινητικότητα των ερευνητών, διότι αυτό αποτελεί σημαντική πύλη για τις χώρες ώστε να οικοδομήσουν αριστεία ε, στον τομέα της έρευνας. Ε, η κινητικότητα αυξάνει κατά πολύ την ποιότητα. Η κινητικότητα είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να προσελκύσει ε, εξαιρετικούς ερευνητές ε, και έτσι να αυξήσει την αριστεία του. Βέβαια, αυτό αποτελεί και απώλεια εγκεφάλων ε, για τους χώρους από τους οποίους φεύγουν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι εάν υπάρχει καλή εισρωή και εκροή ταυτόχρονα, εάν είναι κανείς αρκετά ανοιχτός, μπορεί να προσελκύσει ε, ανθρώπους, μπορεί μάλιστα να επιστρέψουν αυτοί που έχουν διαφύγει. Και μάλιστα συνήθως περισσότερα κερδίζει κανείς από αυτούς που προσέρχονται παρά χάνει από αυτούς που φεύγουν. Ε, είναι λοιπόν μια λύση win-win από την οποία κερδίζουν όλοι. Το ερώτημα είναι λοιπόν πώς θα καταφέρνει η Ευρώπη στη διεθνή αυτή συνεργασία, σε τι, κατά πόσο είναι σε θέση να υποφεληθεί από την πολυπολικότητα. Αν κοιτάξουμε την ε, διεθνή συνεργασία, θα κοιτάξουμε κυρίως ε, τις συνδημοσιεύσεις, τις αποκοινού δημοσιεύσεις. Ε, βλέπουμε πολλές συνεργασίες στον τομέα αυτών στην Ευρώπη. Είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί από ό,τι είναι η Ευρώπη. Οι περισσότερες όμως από αυτές τις συνδημοσιεύσεις είναι ενδοευρωπαϊκές. Έχουμε λοιπόν μια εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά έρευνας ε, και οι περισσότερες διεθνείς ε, συνεργασίες είναι μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να εξετάσουμε και την εξωευρωπαϊκή διάσταση, διότι βλέπουμε ότι ε, οι δημοσιεύσεις Οι συνδημοσιεύσεις Ευρωπαίων με τρίτους ε, διαβάζονται πολύ περισσότερο. από ότι οι καθαρά ευρωπαϊκές. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα αύξησης ε, της επιστημονικής ποιότητας ε, στην Ευρώπη. Αν ε, κοιτάξουμε με ποιους συνεργαζόμαστε και πόσο δραστήριοι είμαστε στις ε, δημοσίευσεις εκτός Ευρώπης, βλέπουμε ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό κόμβο Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών αυτών. Στην επιστήμη λοιπόν υπάρχει πολύ στενός σύνδεσμος, ο οποίος ε, βελτιώνεται συνεχώς. Οι συνεργασίες ε, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αναπτύσσονται πολύ περισσότερο από ότι οι σχέσεις μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οι κυριότερες ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία, έχουν πολύ λιγότερες τέτοιες συνεργασίες. Υπάρχει λοιπόν σημαντικό, σημαντικό υπάρχουν πολύ σημαντικέ δυνατότητε να εκμεταλλευτούν οι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση στι διεθνεί συνεργασίε. και ιδιαίτερα εφόσον γνωρίζουμε ότι αυτού του είδους οι συνεργασίες είναι πολύ πιο πιθανό να οδηγήσουν σε αριστεία. Εάν κοιτάξουμε τις διάφορες χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο ε, συνεργάζεται με τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Κίνα. Ο δεύτερος ε, σημαντικός μηχανισμός είναι η κινητικότητα του, των ε, διεθνών εγκεφάλων. Θα ήθελα και πάλι να σας παρουσιάσω απλά τα βασικά συμπεράσματα. Βλέπουμε και πάλι ότι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη στο θέμα αυτό από ότι ε, η Ευρώπη. Αν κοιτάξουμε πώς κάνουν διδακτορικό, το μεγαλύτερο παραπάνω από το 1 τρίτο στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, είναι αλλοδαπή και μάλιστα πάνω από το 1 τέταρτο προέρχονται από την Κίνα. Και αυτό δεν ε, έχει αλλάξει. Αν το θέτει, βλέπουμε αύξηση. Ε, αντιστρόφως βλέπουμε και ανθρώπου που επιστρέφουν ε, από την Κίνα που το 90% παραμένει στις Ηνωμένε Πολιτείε ακόμα και 10 χρόνια μετά το διδακτορικό τους. Έτσι λοιπόν εποφελούνται οι Ηνωμένε Πολιτείε από τους ε, σπουδαστές αυτές που παραμένουν στη χώρα. Αυτό αποτελεί όφελος και για τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Κίνα. Είναι μια κατάσταση win-win. Ε, αν και μάλλον αυτή τη στιγμή πιο πολύ αποφελούνται οι Ηνωμένε Πολιτείες για τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια πολύ ισχυρή επιστημονική βάση και ότι μπορεί να προσελκύσει τα καλύτερα μυαλά και οι άνθρωποι αυτοί είναι ακόμη καλύτεροι ε, από τους ε, εγχώριους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν τα καλύτερα μυαλά από το εξωτερικό. Η αύξηση λοιπόν σε ποιότητα είναι κατά 12% ε, παραπάνω από ότι το εγχώριο δυναμικό και το μεγαλύτερο μέρος του δυναμικού αυτού ε, προέρχεται από την Κίνα. Είναι βέβαια και πολλοί αυτοί που εγκαταλείπουν τη χώρα. Ακόμα όμως και αν ε, είναι χαμηλότερης ποιότητας από τους ε, εγχώριους επιστήμονες και πάλι βλέπουμε ότι προσελκύουν ε, άλλους ανθρώπους. Ε, έτσι λοιπόν, εάν είναι κανείς ανοιχτός απέναντι στους ανθρώπους που εγκαταλείπουν στις ΗΠΑ, πάλι κερδίζει. Η Κίνα είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικός χορηγός, να το πούμε έτσι, προς τις Ηνωμένε Πολιτείε και χάνουν ε, ε, προσωπικό πολύ, πολύ ποιότητα. ποιότητας. Δηλαδή η Κίνα εξάγει το, τους καλύτερους ανθρώπους ε, που καταλήγουν στις Ηνωμένε Πολιτείε. Έχουμε λοιπόν απώλεια εγκεφάλων για την Κίνα Παρότι όμως οι άνθρωποι που προσέρχονται στην Κίνα ε, είναι χαμηλότερες ποιότητες από αυτούς που εγκαταλείπουν την Κίνα και πάλι είναι υψηλότερο πέτο από αυτούς που βρίσκονται στη χώρα, οπότε και πάλι κερδίζει η Κίνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι και οι δύο πλευρές κερδίζουν και το γεγονός ότι η Κίνα στέλνει τα καλύτερα μυαλά της σημαίνει ότι και πάλι υπάρχει ευκαιρία για την Ευρώπη όχι μόνο να προσελκύσει αυτούς που επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αυτούς που φεύγουν από την Κίνα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το να είμαστε ανοιχτοί. Εντός της Ευρώπης, η πιο Ανοιχτέ χώρες είναι η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βόρεια Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν στενή σχέση ανάμεσα στην αριστεία και το πόσο ανοιχτός είναι κάνει Οι χώρε με τη μεγαλύτερη αριστεία είναι και οι πιο ανοιχτές. Προσελκύουν ε, πολλά ε, ξένα μυαλά τα οποία είναι υψηλότερης ποιότητας από τους ε, ανθρώπους ε, που ήδη βρίσκονται στη χώρα. Είναι όμως πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι από αυτές τις χώρες έχουμε και μεγάλο αριθμό ανθρώπων που εγκαταλείπουν τις χώρες. Δηλαδή και από την Ελβετία και από το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγουν πάρα πολλοί άνθρωποι πολύ υψηλού επίπεδου. Έχουμε λοιπόν, λοιπόν και εδώ πέρα απώλεια εγκεφάλων, αλλά ε, πέρα από brain drain υπάρχει και brain gain, διότι τελικά αυτοί που προσελκύουν ε, είναι καλύτεροι από αυτούς που χάνουν. Πρόκειται λοιπόν για χώρες ανοιχτές, αλλά ανοιχτές ε, και για ανθρώπους που έρχονται, αλλά και για αυτούς που θέλουν να καταλήψουν τις χώρες. Για την Ευρώπη γενικά βλέπουμε σημαντικό brain drain, απώλεια εγκεφάλων, χάνουμε πολλούς εξαιρετικούς ανθρώπους και αυτοί που επιστρέφουν ή αυτοί που έρχονται από άλλες χώρες ε, έχουν πράγματι πολύ υψηλό επίπεδο, δυστυχώς όμως. Αυτοί που έρχονται ή επιστρέφουν ε, είναι ε, λιγότεροι, οπότε το τελικό αποτέλεσμα πράγματι είναι διαφυγή εγκεφάλων. Αυτά λοιπόν γενικά όσον αφορά τη θέση της Ευρώπης, ε, όσον αφορά την αριστεία στην έρευνα. Το επόμενο ερώτημα που εξετάσαμε ήταν το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς έχει συμβάλει σε όλα αυτά. Έχουμε αύξηση στον προϋπολογισμό, αυτό βέβαια είναι πολύ καλό. Ο προϋπολογισμός επικεντρώνεται πολύ συγκεκριμένα στην αριστεία, στην έρευνα και Υπάρχει και ειδικό εργαλείο που επικεντρώνεται στην ε, άριστη έρευνα. Πολύ θετικό λοιπόν το ότι έχουμε αύξηση στον προϋπολογισμό. Ε, βλέπουμε ότι οι επιστημονικές δημοσχεύσεις ε, από το πρόγραμμα αυτό είναι υψηλής ποιότητας. Ε, υψηλότερης ποιότητα από τον διεθνή μεσόωρο, αλλά και γενικά από το τι βλέπουμε στη χώρα αυτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα αυτό αυξάνει την ε, μέση ποιότητα των δημοσιεύσεων, μάλιστα κατά κατά ή τέσσερις φορές σε σχέση με το μέσο όρο. Και για τις, ε, τα 13 παλαιά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμη υψηλότερο το ποσοστό αυτό. το ERC στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. Στόχο έχει ακριβώς να αυξήσει την άριστη έρευνα στις χώρες αυτές. Το άλλο που εξετάσαμε είναι το πρόγραμμα πλαίσιο πώς μπορεί να οδηγήσει σε διεθνείς συνεργασίες και στην διεθνή κινητικότητα ε, διότι αυτό είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της πολυπολικότητας που συζητάμε. Υπάρχει κίνητρο μέσω του προγράμματος ώστε να αυξηθούν οι ενδοευρωπαϊκές συνεργασίες και αυτό εξηγεί και την υψηλή ποιότητα των δημοσιεύσεων σε σχέση με τον μη επιχορηγούμενο δημοσιεύσεων. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των συνεργασιών παραμένει ενδοευρωπαϊκή και έχουμε πολύ λίγες ε, εξωευρωπαϊκές συνεργασίες. υπάρχει ο κίνδυνος ε, να αποθαρρύνεται ο εξω... να αποθαρρύνονται οι εξωευρωπαϊκές συνεργασίες που όμως έχουν υψηλότερη ποιότητα από τις ενδοευρωπαϊκές συνεργασίες. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο βελτίωσης του προγράμματος πλαισίου ώστε να βελτιωθούν και οι εξωευρωπαϊκές συνεργασίες. Ο δεύτερος σημαντικός μηχανισμός είναι η διεθνής κινητικότητα ε, των αρίστων και έχουμε για παράδειγμα το πρόγραμμα Marie Curie και όλα τα άλλα προγράμματα μπορούν να ενθαρρύνουν την κινητικότητα, αλλά αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο και στοχευμένο εργαλείο και ε, αυτές ε, οι υποτροφίες ε, χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για διδακτορικά, αλλά αυτές οι υποτροφίες ενθαρρύνουν την κινητικότητα. Οι περισσότερες υποτροφίες αυτές, λοιπόν, δαπανώνται σε μεγάλο βαθμό εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελάχιστοι πόροι χρησιμοποιούνται για συνεργασίε με τις ΗΠΑ, Πολιτείες, ενώ έχουμε πολύ μικρή εκπροσώπηση τη Κίνας. Οι υποτροφίες αυτές μπορούν να, να, βοηθ... μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βοηθήσουμε και όσους επιστρέφουν αλλά γενικά οι βελτιώσεις αυτές αφορούν πολύ μικρό κομμάτι του προγράμματος, ε, το οποίο γενικά αποτελεί πύλη για βελτίωση της κατάστασης. Ποιες είναι λοιπόν οι συστάσεις μας για την ε, μελλοντική πολιτική. Νομίζω ότι είναι ήδη σαφή αυτά από αυτά που ήδη συζητάμε. Το θέμα είναι ε, πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον. το, το τοπίο τεχνολογίας και επιστήμης ε, θα παραμείνει ανοιχτό και διασυνδεδεμένο. Αυτό είναι άγνωστο, όλα είναι πιθανά. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ πιο σωστρεφή αντιμετώπιση. Πάντως ε, σημαντικό είναι ότι για την άριστη έρευνα σημαντικό είναι να διατηρήσουμε ένα παγκόσμιο τοπίο ανοιχτό και διασυνδεδεμένο. Ακόμη όμως και αν ε, αποσυνδεθούν ε, μεταξύ τους οι πόλοι αυτοί, ποια θα πρέπει να είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κίνα αποτελεί ήδη αρκετά σημαντικό πόλο ώστε να μπορεί να επιβιώσει μόνη της. Ε, θα συνεχίσει να επωφελείται από το να είναι ανοιχτή, αλλά θα μπορούσε να επιβιώσει και μόνη της. Οι Ηνωμένε Πολιτείες εξαρτώνται από την προσέλκυση ε, εγκεφάλων και έτσι θα ε, έχανε την ε, θέση της, ίσως όχι αρχικά, αλλά σε βάθος χρόνου θα αρχίσει να χάνει τη θέση της. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι τέτοιο θα είναι βιώσιμο μόνο εάν αποτελέσει έναν ενωμένο πόλο, έναν ενιαίο πόλο, διότι σημαντικό εδώ είναι το μέγεθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πιο σημαντικές συστάσεις μας λοιπόν είναι ότι χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, να ε, ε, έχουμε επαφές μαζί τους ε, και να επενδύσουμε στην αριστεία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Θα πρέπει δηλαδή να διατηρήσουμε την αριστεία, διότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προσελκύσουμε άλλους. Αυτό απαιτεί συνεχή δέσμευση ε, για μια εσωτερική ενιαία αγορά έρευνας. Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε και ε, τον υπόλοιπο κόσμο. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, να μπορούμε να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε να ε, στείλουμε αρίστους ή να προσελκύσουμε αρίστους από άλλα μέρη του κόσμου. Αυτή λοιπόν είναι η βασική μου πρόταση. Θα ήθελα να κλείσω εδώ και περιμένω να ακούσω τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας. Σας ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εφόσον ξεκινήσαμε αργά, θα σας ζητήσω να σεβαστείτε το χρόνο. Να ξεκινήσουμε από τους συντονιστές. Έχετε δύο λεπτά ακριβώς. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε, κύρια Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά που έχουμε κοντά μας την ομιλήτρια. Έχουμε δουλέψει μαζί εδώ και για πολλά χρόνια. Την καλωσορίζουμε λοιπόν στην Επιτροπή Ήτρε. Έχω δύο σχόλια, παύλα ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει συνεργατική έρευνα από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά η, η έρευνα. Δώσατε έμφαση στην συνεργασία. Και ξέρουμε ότι το πρόβλημα ήταν πάντοτε το, το πλαίσιο, πώς θα δημιουργηθεί δηλαδή αυτός ο χώρος συνεργασίας εντός της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την έρευνα. Αρκετά κοινά άρθρα έχουν δημοσιευθεί χάρη σε αυτά τα προγράμματα πλαίσια. Μάθαμε πώς να συνεργαζόμαστε στην έρευνα και υπάρχει τώρα η τάση να βασιζόμαστε όλο και περισσότερο σε μεμονωμένες ομάδες που ασχολούνται με την καινοτομία. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το κατά πόσο είμαστε ανοιχτοί στην, στην έρευνα στο ζήτημα της καινοτομίας. Έχω την τάση να σκέφτομαι ότι η επιστήμη θα πρέπει να είναι ανοιχτή στον κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ η καινοτομία είναι κάτι πιο τοπικό, είναι ένα φαινόμενο ε, περιφερειακό. Η συνεργασία όμως και αυτό το άνοιγμα στην έρευνα είναι σε πολλές περιπτώσεις πιο δύσκολο. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθείτε λίγο σε αυτό το ζήτημα του κατά πόσο μπορεί να είναι ανοιχτή η καινοτομία σε ό,τι αφορά την έρευνα και την επιστήμη. Ευχαριστούμε πολύ. Από το S&D υπάρχει κάποιος που να θέλει να πάρει το λόγο. Όχι, αν όχι, κυρία Ταλαμπάιοβα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη. Δύο σύντομες ερωτήσεις μόνο. Πρώτα απ' όλα, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ούτω ώστε να προσελκύσουμε περισσότερους επενδυτές, να μπορέσουμε να συνδυάσουμε επενδύσεις και ε, δημόσιες χρηματοδοτήσεις στον τομέα της έρευνας. Το δεύτερο σημείο, αν πιστεύετε εσείς μετά τα πορίσματα της έρευνάς σας η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί ορθά όλες τις συνεργίες, για παράδειγμα μεταξύ της έρευνας και της εκπαίδευσης και της συνεργίες χρηματοδότησης. Περιφερειακά εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Ε, στην αρχή αναφερθήκατε σε κάποια ενδιαφέροντα πορίσματα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Ποια είναι η βάση για αυτή τη συνεργασία, μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένοι. Και το τελευταίο μου ερώτημα είναι ίσως λίγο πιο φιλοσοφικό. Τι μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη για να κρατήσουμε αλλά και να προσελκύσουμε νέους ερευνητές, νέες ηλικίε. Πώς μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Είναι καλύτερα να εκπαιδεύσουμε μια νέα γενιά ή να προσελκύσουμε εγκεφάλους από ολόκληρο τον κόσμο. Πώς μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί εγώ φοβάμαι ότι στην Ευρώπη θα λείψουν αυτά τα σπάνια ταλέντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νινής το έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Είναι ιδιαίτερα σημαντική και είναι και πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο ανταγωνισμό με την Κίνα και τις Ηνωμένε Πολιτείες στον τομέα της έρευνας και της α, τεχνολογικής ανάπτυξης. Ως Φινλανδός, για μας στη Βόρεια Ευρώπη, ε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών είναι πολύ σημαντική και είναι ενδιαφέρον ότι το, το βρήκατε κι εσείς στην ε, έρευνά σας. Όχι μόνο στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η συνεργασία σε ολόκληρο τον κόσμο είναι σημαντική για την επιτυχία της ε, έρευνας. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε το ότι η επιστημονική κοινότητα είναι ανοιχτή σε συνεργασία και αν έχετε να πείτε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό θα ήμουν ευτυχής να το ακούσω. Έχω τρία ακόμη σχόλια που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Το ένα έχει να κάνει με τις δαπάνες για την έρευνα. Αν ρίξετε μια ματιά στο τι ξοδεύουν στην Κίνα για την έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και στην Νότια Κορέα, οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη δεν αυξάνουν τον προϋπολογισμό τους και κυρίως σε επίπεδο κρατών μελών. Τι θα πρέπει να κάνουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη. Ε, αναλογικά με το, με το GDP της κάθε χώρας. Το άλλο σχόλιο έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε επιστήμονες και να τους κρατήσουμε εδώ στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό για μας να προσελκύσουμε επιστήμονες, όχι μόνο από το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται πολύ καλή υποδομή πώς μπορούμε μακροπρόθεσμα να εφαρμόσουμε μια στρατηγική για την έρευνα και τις υποδομές, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι ενδιαφέρον και για τους ερευνητές να έρθουν σε εμά στην Ευρώπη. Και το τρίτο σημείο έχει να κάνει με το πόσο μπορεί να είναι ανοιχτή η έρευνα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την κινητικότητα, αλλά και σε ό,τι αφορά τα δεδομένα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα, ας πούμε, μια βάση δεδομένων που να είναι ανοιχτή και να προωθεί αυτού του τύπου την ε, πρόσβαση για όλους τους ερευνητές. Σας Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόρκια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την εκπόνηση της μελέτης και ευχαριστώ και για την ε, σημερινή παρουσίαση. Θέλω να σας ρωτήσω, σε σχέση με την ε, απορρόφηση ταλέντων από τρίτες χώρες, ποιοι είναι οι τομείς που πιστεύετε πως θα υπήρχε ανάγκη από εξωτερική συμβολή, ώστε ακριβώς να σημειωθεί πρόοδο σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Επιπλέον, ε, Έχουμε αναλύσει το πρόβλημα της φυγής εγκεφάλων από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Ε, από τη μια πλευρά ε, πρόκειται για κάτι το οποίο αποτελεί τεράστια ευκαιρία για τους ερευνητές, αλλά από την άλλη στην ουσία φτωχαίνουν τα εθνικά ερευνητικά τμήματα. Πέρα από την αύξηση του προπολογισμού υπάρχουν λύσει στις οποίες θα μπορούσαμε να στραφούμε για να, για να αναχαιτήσουμε αυτό το πρόβλημα. Και έπειτα μια διευκρίνηση. Ποιοι είναι οι παράγοντες που περιορίζουν τον θετικό αντίκτυπο των ερευνητών που επιστρέφουν στις χώρες τους και κατά τη γνώμη σας ποια είναι τα εμπόδια και πώς θα μπορούσαμε να τα άρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλοι συντονιστές, να δώσουμε το λόγο στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ποιο θέλει να πάρει το λόγο. Uh, Για ένα λεπτό έχετε στη διάθεσή σας. Πρώτα απ' όλα κυρία Μαρκές. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και για την ε, εισήγησή σας. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με την αριστεία και το να μην μένουν πίσω κάποιο, ε, κάποιοι ερευνητές. Ήδη σήμερα το πρωί συζητήσαμε πώς θα μπορούσαμε, χωρίς να, χωρίς καταλήψουμε το κριτήριο της αριστείας, να είμαστε πιο... Ε, δεκτική εντός της Ευρωπαϊκή Ένωσης και τώρα σε σχέση με τις τρίτες χώρες το πρόβλημα μας είναι να ε, προσελκύσουμε τα ταλέντα ε, προφανώς εκεί υπάρχει πρόβλημα αλλά επίσης ε, το θέμα είναι να σκεφτούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε τη συνεργασία με τρίτες χώρες και όχι μόνο με τους ανταγωνιστές μας την Κίνα και τη ΣΥΠΑ δηλαδή αλλά και άλλες χώρες όπου μπορούμε να αναπτύξουμε ταλέντα αλλά και να τα αφήσουμε εκεί όπου βρίσκονται, όχι απαραίτητα να τα φέρουμε εδώ το ταλέντο, να αναπτυχθεί το ταλέντο μέσω της ισότιμης συνεργασίας ανάμεσα στα δικά μας ερευνητικά κέντρα και τα ερευνητικά κέντρα τρίτων χωρών και όλος ιδιαίτερος σε υπήρους πιο ξεχασμένες όπως είναι η Αφρική. Σας ευχαριστώ πολύ ε, για την απάντησή σας και των προτέρων. Σας ευχαριστώ και εγώ. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Η ομιλήτρια είναι εκτός μικροφώνου. Με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Σε σχέση με την παγκόσμια επιστήμη, υπάρχει συνένεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λειτουργεί ως ένα μπλοκ. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο προωθεί κυρίως τον ανταγωνισμό με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι την συνεργασία από ό,τι βιδάμε και στην έρευνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ευνοήσει την εσωτερική συνεργασία και όχι τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Σε ό,τι αφορά τώρα την κινητικότητα, κάναμε λόγο για, για το λεγόμενο brain drain, για την φυγή εγκεφάλων. Έχουμε δηλαδή τα εγχώρια ταλέντα που φεύγουν. Υπάρχει όμως και άλλος τρόπος, ο πιο τεμπέλικος θα λέγαμε. Θα μπορούσαμε δηλαδή να εισάγουμε Κινέζους, για παράδειγμα, κατόχους διδακτορικών διπλωμάτων, να δουλέψουν σε διάφορα πανεπιστήμια και να μοιραστούν ε, τις γνώσεις τους, αντί να εκπαιδεύσουμε τους δικούς μας. Αυτό λοιπόν που ανησυχώ εγώ είναι ότι μπορεί να θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένας παγκόσμιος παίκτη ό,τι αφορά την έρευνα και την επιστήμη, αλλά τελικά καταλήγει να είναι ένα σύστημα πολύ κλειστό. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποιο άλλος. Αν όχι, να δώσουμε πίσω το λόγο στην ε, ομιλητριά μας για να δώσει απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα ερωτήματα. Είναι εξαιρετικά ερωτήματα. Αυτά είναι, αυτά που συζητήσατε εσείς εδώ, είμαι σίγουρη, με κάνουν να πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο κάνει εξαιρετική δουλειά. Επιτρέψτε μου λοιπόν να προσπαθήσω μία-μία να απαντήσω στις ερωτήσεις σας με τη Μαρία Γράσια να ξεκινήσουμε σε ό,τι αφορά τα προγράμματα συνεργασίας. Πώς αυτό συμβαδίζει με τις μεμονωμένες ομάδες. Αυτό που βλέπουμε είναι όντως να ενδιαναμώνονται οι ομάδες. Πολλές από τις ομάδες αυτές είναι ιδιαίτερα διεθνείς. Επομένως έχουμε την ίδια στιγμή κινητικότητα ταλέντων αλλά και συνεργασία πολύ συχνά έχουμε διεθνή συνεργασία η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι στην ίδια ομάδα έχεις άτομα που προέρχονται από διαφορετικούς οργανισμούς. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν οι μεμονωμένες ομάδες και η συνεργασία λειτουργούν ταυτόχρονα μια χαρά. Αν οι ομάδες αυτές είναι από μόνες τους αρκετά ανοιχτέ σε ό,τι αφορά την κινητικότητα κτλ. Δεν θεωρώ λοιπόν εγώ ότι το, το ένα αποκλείει το άλλο, θεωρώ ότι το ένα ενδυναμώνει το άλλο. Έχουμε διεθνή κινητικότητα και συνεργασία. Από κοινού ενδυναμώνουν ε, το μηχανισμό αυτόν. Κάποιοι επίσης παρατήρησαν αυτή την ιδέα της ανοιχτής κοινότητας στην επιστήμη. Είναι πιο εύκολο να το καταλάβουμε όταν μιλάμε για καινοτομία. Είναι αλήθεια ότι όσο πιο πολύ προσεγγίζουμε την εμπορευματική χρήση, τόσο πιο δύσκολο είναι να έχουμε αυτή την κατάσταση win-win, γιατί είναι σημαντικό κάποιος να είναι καλύτερος από τους ανταγωνιστές του. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι Υπάρχουν πολλές συνεργασίες σε ό,τι αφορά την καινοτομία. Αρκετές εταιρείες συνεργάζονται μεταξύ τους από διάφορες χώρες. Σε πολλές περιπτώσεις οι χώρες αυτές που έχουν ιδιαίτερα έντονες συνεργασίες, διεθνείς συνεργασίες, αλλά και μεγάλη κινητικότητα. Αν δηλαδή προσελκύεις πολλά ταλέντα, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα παραμείνουν στον ακαδημαϊκό χώρο, θα μετακινηθούν σε διάφορες εταιρείε και εκεί θα δημιουργήσουν με τη σειρά τους διάφορους διεθνείς συνδέσμους. Επομένως, έχεις αυτή την, ε, το, το, το, την τεράστια βάση δεδομένων διεθνών ταλέντων και μπορείς να χρησιμοποιήσεις την παγκοσμιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επό αυτήν την έννοια, λοιπόν, αυτή η έλλειψη συνόρων, αν θέλετε, στην επιστήμη είναι κάτι το οποίο λειτουργεί καλά. Και οι εταιρείε μπορούν να προσελκύσουν αυτούς τους ερευνητές και να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα αυτής της παγκοσμιοποιημένης επιστήμης. Μια άλλη καλή ερώτηση ήταν κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί όσο πρέπει τις συνεργίες μεταξύ των διαφόρων οργανισμών αλλά και μεταξύ των εθνικών επιχορηγήσεων και των προγραμμάτων πλαισίων. Σίγουρα στα πλαίσια των προγραμμάτων πλαισίων θα μπορούσαν να υπάρξουν πολλές περισσότερες συνεργίες που να εκμεταλλευόμαστε. Εγώ αναφέρθηκα απλά στην ε, επιχορήγηση Marie Curie ως επιχορήγηση κινητικότητας αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει καλά με το όργανο για τη συνεργασία. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω πιστεύω ότι είναι σαφέ ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα πλέον αν κανείς επωφεληθεί στο δυνατόν περισσότερο από τις συνεργίες αυτές. Παρ' όλα αυτά όμως όταν υπάρχουν και τοπικές επιχορηγήσεις όπου βρίσκονται αυτές οι συνεργασίες, αυτοί οι ερευνητές, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται και οι πόροι αυτοί, ούτως ώστε να χτίζεται και τοπική υποδομή, ούτως ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν τα ταλέντα αυτά ερευνητές αυτοί όταν επιστρέψουν. Κυρίως για αυτές τις χώρες που θα μπορούσαν να υποφεληθούν πολύ περισσότερο προσελκύοντας και ξένους ερευνητές, ξένα ταλέντα πώς να προσελκύσουμε ταλέντα ερευνητέ, αυτό είναι ένα ερώτημα που έχει προκύψει πολλές φορές. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι προσελκύουμε ταλέντα. Έχουμε, υπάρχει κάποια ανάλυση σε επίπεδο δεδομένων όπου αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που κάνει κάποιον να, να θέλει μεγαλύτερη κινητικότητα σε διεθνές επίπεδο, αν υπάρχει βέλερ μέσω των προγραμμάτων πλαισίων, αυτό που είναι πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μετακίνηση, που συνήθως είναι ιδιαίτερα ταλαντούχοι, ο λόγος που μετακινούνται είναι γιατί τους βοηθάει στην καριέρα τους σε ό,τι αφορά την έρευνα. Το να μπορούν δηλαδή να λειτουργούν πάντα σε επίπεδο εχμής, να είναι όσο το δυνατόν πιο προηγμένη η έρευνά τους. Γι' αυτό λοιπόν και θέλουν να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ερευνητικής αριστείας. Εδώ είναι το, το σημείο κλειδί ερευνητική αριστεία και η δυνατότητα να συνεργαστούν με άλλους ερευνητές ε, ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Επομένως η συνδεσιμότητα αυτή και η έλλειψη συνόρων, το άνοιγμα των συνόρων είναι εξαιρετική παράγοντες για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερα ταλέντα. Αυτό είναι που ψάχνουν οι ερευνητέ που μετακινούνται, τα ταλέντα που μετακινούνται. Άλλα ερωτήματα για την διεθνή και τοπική συνεργασία και επίση το ερώτημα για την συνεργασία στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δύο αυτά σημεία πιστεύω ότι είναι αλληλοσυμπληρωματικά. Δεν νομίζω ότι το ένα μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο. Έχουμε τοπική συνεργασία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να χτίσουμε αριστεία. Αλλά ποτέ δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τη συνεργασία με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, όταν έχουμε μια σταθερή συνεργασία σε εσωτερικό επίπεδο, τότε θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως δέλεαρ για ακόμη περισσότερη συνεργασία, για καλύτερη συνεργασία με ε, εταίρους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ε, θα πρέπει ποτέ να το αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίζουμε αυτό ως δίλημα ή το ένα ή το άλλο. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε την επιστημονική έρευνα με εσωτερική συνεργασία και στη συνέχεια να υποφεληθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο με εξωτερική συνεργασία. Το ένα συμπληρώνει το άλλο όπως βλέπετε. Τι άλλο έχω εδώ πρόσβαση στην υποδομή, υποδομή έρευνας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους ερευνητές που μετακινούνται. Η δυνατότητα δηλαδή να έχουν την τελευταία υποδομή, όχι μόνο υποδομή, οποιονδήποτε τύπου, α, οποιοδήποτε τύπου εξοπλισμό αυτό ενδιαφέρει και τα εγχώρια ταλέντα, τους εγχώριους α, ερευνητές. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να προσελκύσει το ενδιαφέρον. Επομένως, χρηματοδότηση της ε, υποδομής είτε με τις επιχορηγήσεις Marie είτε με άλλες επιχορηγήσεις και πάλι θα είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να υποφεληθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε πολλές περιπτώσεις αναφέρθηκε το ζήτημα της διαρροής εγκεφάλων, κυρίως για τον νότο. Ποια είναι η λύση για αυτή τη φύγη, για τη διαρροή εγκεφάλων. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ε, να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη φυγή εγκεφάλων απλά σταματώντας την, την εκροή ερευνητών η διαρροή εγκεφάλων, πώς να λύσεις αυτό το πρόβλημα, μα να εξασφαλίσεις ότι μπορούμε να τους στείλουμε πίσω όλους αυτούς τους ερευνητές, αλλά να ξέρουμε ότι θα επιστρέψουμε και να δουλεύουν σε πλαίσια ανοιχτών συνόρων. Να φροντίσουμε να επιστρέψουν και βεβαίως να μπορέσουμε να εξαφανίσουμε τα εμπόδια όλα αυτά που δεν τους επιτρέπουν να επιστρέψουν, να επιστρέφουν στις χώρες τους. Είναι βέβαιο ότι θα επιστρέψουν στις χώρες τους αν δεν θεωρούν ότι βάζουν σε κίνδυνο τις ερευνητικές τους καριέρες. Επομένως πρέπει να έχουμε δυνατά τοπικά συστήματα έρευνας, όχι μόνο σε κάθε χώρα. Και πάλι θεωρώ ότι θα πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, θα πρέπει να εξετάζουμε το ερευνητικό περιβάλλον ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως και πάλι να μπορούμε να κρατάμε ανοιχτά τα, τα, ερευνητικά σύνορα είναι ένας τρόπος να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αρκετούς ερευνητές, αρκετά ταλέντα που θα θέλουν να επιστρέψουν. Και περνάμε τώρα και αυτό το, το σημείο, πώς μπορούμε να έχουμε συνοχή και αριστεία αλλά και συμπερίληψη. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να εξακολουθήσουμε να δίνουμε έμφαση στο γεγονός ότι όλοι αυτοί οι ερευνητές έχουν στόχο να χτίσουν την αριστεία και αν θέλουμε να έχουμε αριστεία τότε θα πρέπει να έχουμε και κινητικότητα. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει και συμπερίληψη, ότι υπάρχει και συνοχή όμω Αυτά τα σημεία όλα δεν υποκαθιστούν το ένα το άλλο, δεν αντικρούν το ένα το άλλο. Αν θέλουμε να έχουμε συμπερίληψη, αν θέλουμε να έχουμε συνοχή, τότε θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτήν την ε, κατάργηση των επιστημονικών συνόρων, τόσο ώστε να μπορέσουμε να χτίσουμε αριστεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τελευταίο σημείο που έχω σημειώσει, υπάρχει ένα πιο ε, τεμπέλικο, πιο εύκολος ε, τρόπο. δηλαδή να προσελκύσουμε για παράδειγμα Κινέζους αντί να εκπαιδεύσουμε τους δικούς μας ερευνητές. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέτοια εύκολη λύση, δεν υπάρχει τέτοια τεμπέλικη προσέγγιση. Οι καλύτεροι των Κινέζων ερευνητών θα έρθουν μόνο στα ερευνητικά περιβάλλοντα που θα είναι άριστα, που θα είναι τα καλύτερα δυνατά. Επομένως, αν δεν επενδύσουμε σε μια τοπική επιστημονική βάση, σε, σε μια εκπαίδευση ερευνητών, οι καλύτεροι Κινέζοι δεν, δεν θα έρθουν. Επομένω, ο μόνο τρόπο να, του, ο μόνος τρόπος να του προσελκύσουμε και όλου αυτού του ερευνητέ από του οποίου θα μπορούσαμε να υποφεληθούμε δηλαδή, είναι επενδύοντα εμεί οι ίδιοι και επενδύοντα στην, στην αριστεία πρώτα απ' όλα εμεί. Σα ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό και η παρουσίασή σας ε, πολύ ε, σημαντική και πολύ ενδιαφέρον το θέμα για μας και κυρίως εν ώψη του επόμενου προγράμματος πλαισίου. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Είμαστε βέβαιοι ότι θα το ξανασυζητήσουμε. Είστε εμπειρογνώμονας επί του θέματος. Σας ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε. Uh, τώρα, συνάδελφοι, τώρα πρέπει να μιλήσουμε για τον κύριο Λέπαρ που είναι ο, επόμενο, που είναι ο νεοεκλεγής υποψήφιος για το τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια, της ΕΝΙΖΑ. Καλωσορίσατε. Να σας θυμίσω το άρθρο 36 από το ε, του ε, κανονισμού της ΕΝΙΖΑ ε, που ορίζει ότι πριν να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ο εκτελεστικός διευθυντής καλείται να ε, έρθει σε συνέντευξη με το Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό έχουμε σήμερα προγραμματίσει μία ώρα ε, συνομιλία μαζί σας. Θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να σας ρωτήσουμε ερωτήσεις, ε, να ρωτήσετε κι εσείς και να σας απαντήσουμε. Ελπίζουμε πώς θα είναι καρποφόρα η σημερινή μας συζήτηση. Έχετε λοιπόν το λόγο κύριε Λεπασάρα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ε, σας συστηθώ και να συζητήσουμε μαζί τι μπορεί να κάνει η ΕΝΙΣΑ για να βελτιώσει το επίπεδο της κυβερνοασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο μια τεχνική ε, πρόκληση με την οποία ασχολούνται οι ειδικοί της πληροφορικής, αλλά αποτελεί και μια πολιτική και κοινωνική πρόκληση. Το νέο νόμος για την κυβερνοασφάλεια θεωρεί ότι είναι αυτή η ραχοκοκαλιά της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, εσωτερικής αγοράς που είναι πολύ σημαντική για τη ζωή μας, που καθοδηγεί την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσπίζει την κυβερνοασφάλεια ως ένα τομέα που στηρίζει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων επιγραμμικά σε τομείς κλειδιά όπως η τηλεπικοινωνία, η οικονομία, οι μεταφορές και πολλοί άλλοι πέρα από τις ε, εθνικές και τις ε, ενωσιακές στρατηγικές ε, όσον αφορά το επιγραμμικό περιβάλλον, αυτό απαιτεί την εμπειρογνωμοσύνη και ειδικότητε που μπορούν να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Μεγάλες προσδοκίες λοιπόν για την ε, κοινότητα κυβερνοασφάλειας. Η ΕΝΙΖΑ έχει την αποστολή να συμβάλλει στην επίτευξη ενός υψηλού επίπεδου ε, κυβερνοασφάλειας ολόκληρη την Ένωση. Έχει αναπτυχθεί ως ένας κόμβος εμπειρογνωμοσύνης για την κυβερνοασφάλεια και ε, ως και μάλλον και έχει αναλάβει έναν ε, ρόλο διευκόλυνσης. Ε, και τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν όντω αυξηθεί οι δυνατότητε τη ΕΝΙΖΑ. Μέσα στο σημερινό πλαίσιο που η κυβερνοασφάλεια έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε όλου του πολιτικού τομεί και τα επίπεδα τη κοινωνία και όπου οι προκλήσει είναι πολύπλευρε ε, και πολυσχηδεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οθετήσει ένα συνολικό ε, πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο και η Επιτροπή σας έχει συμβάλει μέσω της ε, γετικής του ηγετικού ρόλου που έπαιξε για την ε, σχετική νομοθεσία. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή Γέζη Μπούζεκ και την καθηγήτρια Αγγέλικα Νίβλερ που ηγήθηκαν τη εργασία για το νόμο περί κυβερνοασφάλεια και όλου του ευρωβουλευτέ που συνέβαλαν στην ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου για την κυβερνοασφάλεια, Όπω η κυρία Πιλάρ Δικαστήγιο για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Τηλεπικοινωνιών, όπου υπάρχουν σημαντικές διατάξεις που αφορούν την ε, κυβερνοασφάλεια. Να ευχαριστήσω το Ευρωκοινοβούλιο που μα δίνει, μα προσέφερε το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Ε, ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει ε, αυτό που έχει αποτελέσει ο σχετικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων και των προσωπικών στοιχείων, δηλαδή τον χρυσό κανόνα εμπιστοσύνης. Όμως τα κρατημέλη μόλις τώρα αρχίζουν να εφαρμόζουν ε, την οδηγία EMIS και είναι πολύ πρόσφατη η ισχύ του. Ε, η υπηρεσία μας όμως έχει ενισχυθεί μέσω της νέας εντολής ώστε να εκμεταλλευτεί πλήρως το νέο πλαίσιο. Μπορεί αυτό να το πράξει βασιζόμενη στις, ε, στα δυνατά της στοιχεία, αλλά και ανταποκρινόμενη στις νέες ανάγκες της Ένωσης μέσω του νέου νομοθετικού πλαισίου. Να σας πω τώρα πώς βλέπω το ρόλο της υπηρεσίας αυτής τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο της ε, ασφάλειας των πληροφοριών αλλά και της, ε, το πλαίσιο της ε, κυβερνοασφάλειας. Στο πλαίσιο της προστασίας των πληροφοριών, η υπηρεσία μας θα πρέπει να συμβάλλει στο πώς καλύτερα θα επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας και πώς θα χειριστεί τους τομείς ε, που περιλαμβάνονται εκεί. Θα πρέπει να προβούμε σε συστηματική ποιοτική ανάλυση της ε, κυβερνοασφάλειας, της προστασίας μάλλον τη πληροφορία στα διάφορα κράτη-μέλη, γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει μέσω της ομάδας συνεργασίας τα κράτη-μέλη να διαδώσουν τις καλές πρακτικές και να βοηθήσει να δημιουργηθεί μια κοινή ε, λογική όσον αφορά την προστασία των ε, πληροφοριών ε, σε συνεργασία με ε, τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές. Επίσης μπορούμε να παρέχουμε αναλύσεις για το πώς καλύτερα θα μπορούσαμε να χειριστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα θέματα κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο του IG και τη μετακίνηση από τις υποδομές στο νέφος. Επίσης μπορεί να βοηθήσει στην δημιουργία δυνατοτήτων θεσπίζοντας και συντηρώντας ένα δίκτυο εμπειρογνωμονών και ε, ε, ειδικοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση από τις οποίες θα μπορεί να αντλήσει την ε, στοχευμένη βοήθεια που θα χρειαστεί ένα περίπτωση. Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε βοήθεια στα κράτη-μέλη για ανθεκτικότητα όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και βασισμένη στη συμβολή ιδιωτικών αλλά και δημοσίων φορέων καθώς και άλλων αρμόδιων δημοσίων ε, ε, υπηρεσιών. Τώρα, μέσα στο πλαίσιο της ΕΝΙΖΑ θα πρέπει να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη ανάμεσα στους φορείς, να αυξηθεί μάλλον η εμπιστοσύνη, να αυξηθεί η συνεργασία, η, επίσης να δημιουργηθούν ομάδες, ε, τομεακές ομάδες άμεσης αντίδρασης σε απειλές, αλλά να γίνονται και κοινέ ασκήσεις, ώστε να δημιουργηθούν δυνατότητες ταυτόχρονης και κοινή απάντησης και ανταπόκρισης σε κινδύνους. Ε, μέσω της γραμματείας μας μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αποκομίσουν διδάγματα από τις εκθέσεις, τις αναφορές περιστατικών. Τέλος, θα πρέπει να συμβάλλουμε στο να βελτιωθεί η ε, γνώση όσον αφορά τα προβλήματα αυτά και να βελτιωθεί και η, υγιεινή ε, ενώ θα ενεργούμε όλοι ε, με τις καλύτερες πρακτικές για να μπορέσουμε να χειριστούμε καλύτερα τους ε, ε, κινδύνους. Έχουμε δε τα παραρτήματα της οδηγίας. Μέσα σε αυτά αναφέρεται η παρότρινση των καλύτερων πρακτικών όσον αφορά την μη αποκάλυψη στοιχείων ο οργανισμός μας θα πρέπει να βοηθήσει την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη στο να θεσπίσουν ένα σαφές επιχειρησιακό σχέδιο όσον αφορά τα ε, σχέδια ε, κοινοποίησης ε, αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της βιομηχανίας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της δημιουργίας δεσμών, μέσω των ισχυών των πλαισίων πιστοποίησης, να σχεδιαστεί ένα διαφανές και ανοιχτό πλαίσιο που θα διέπει την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την πιστοποίηση των σχεδίων αυτόν αυτών ε, πιστοποίησης, έτσι ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια όλων. Θα πρέπει να βασιστούμε στο υπάρχον ε, πλαίσιο δυνατοτήτων ε, και εμπειρογνωμοσύνης, αλλά να αναζητήσει και την εξασφάλιση της ε, ισορρόπησης των ε, διαφόρων ε, συμφερόντων των ενδιαφερειμένων φορέων. Εμείς ερχόμαστε, μάλλον ο οργανισμός ε, ε, έρχεται σε διαβούλευση σε πρώιμο στάδιο για κάθε σχέδιο. Μπορούμε να φτιάξουμε δε ε, δυνατότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως, αλλά και να προωθήσουμε τις προσεγγίσεις εξασφάλισης της προστασίας από το σχεδιασμό ε, των προγραμμάτων. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση επίσης να μεταφράσουμε τις συχνά πολύ τεχνικές γνώσεις σε γνώση και σε γλώσσα κατανοητή για τους μη ειδικού. Και αυτό γιατί χρειάζεται η κυβερνοασφάλεια σε διάφορους τομείς σε ολόκληρη την Ένωση. Αυξάνοντας λοιπόν την ε, ε, ε, λειτουργία μας θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την Ένωση να δημιουργήσει ανθεκτικότητα σε πολλούς τομείς. Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε για το συντονισμό και τη δημιουργία ή αύξηση δυνατοτήτων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που εμπίπτουν στην εντολή μας. Δεν μπορούμε ωστόσο να ε, ανταποκριθούμε σε αυτή την εντολή μόνοι μας. Οι πόροι μας δεν είναι απεριόριστοι. Ε, πρέπει να έρθουμε σε επαφή με πολύ περισσότερους ε, ενδιαφερόμενους φορείς, να οικοδομήσουμε συμμαχίες και να αναπτύξουμε δίκτυα συνεργασίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με διάφορους φορείς, με τα κρατημέλη και με τον ιδιωτικό τομέα. Ο επανεστιασμός του καταλόγου υπηρεσιών της ΕΝΙΖΑ θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στα προγραμματικά έγγραφα του οργανισμού. Ελπίζω πως θα μπορέσω να βοηθήσω το Συμβούλιο να φτάσει σε συμφωνία για ένα σαφές ε, σύνολο επιχειρησιακών στόχων με βάση τις αποστολές του οργανισμού. Είναι σημαντικό ο οργανισμός αυτός να διατηρήσει το καλό σκόρ της όσον αφορά την ε, δημοσιονομική διαχείρισή της. Ε, ε, η ΕΝΙΣΑ είναι ένας οργανισμός που ιστορικά έχει αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τη διατήρηση και ανάπτυξη των ειδικοτήτων και των ταλέντων που χρειάζεται. Πολλές από αυτές τις προκλήσεις αναφέρονται στη τελευταία έκθεση απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης είναι ένας οργανισμός ε, υπομετάβαση με ε, περιορισμένες χρονικά ε, εντολές και αλλαγή έδρας σε αυτό το τομέα θα πρέπει να συνεννοηθούμε με τις ε, ελληνικές αρχές και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις ε, δυνατότητες του οργανισμού μας. Ένα σταθερό, ε, μια σταθερή έδρα και μια ξεκάθαρη εντολή θα ενισχύσουν το ρόλο της Ιουνής. Αλλά αυτά δεν αρκούν, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια κουλτούρα όπου θα ε, μπορούμε να παράγουμε προστιθέμενη αξία και θα βοηθήσουμε στο να αναπτυχθούν σε ολόκληρη την Ένωση φορείς συνεργασίας. Η εθνική ε, εμπειρογνώμονες ε, μέσω της ε, περιοδικής εναλλαγής θα βοηθήσουν στο να δημιουργηθούν δίκτυα συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη ώστε να δημιουργηθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και να αντιμετωπιστεί έλλειψη ειδικοτήτων. Θέλω να σας ευχαριστήσω κλείνοντας για τη στήριξή σας σε αυτήν την, σε αυτήν την υπηρεσία, για το ότι εξασφαλίσατε μια σταθερή εντολή και μια σταθερή νομική βάση. Ελπίζω πως αυτή η αρχική ανταλλαγή απόψεων θα σημάνει την, ε, έναν μόνιμο διάλογο ανάμεσα στον οργανισμό και το Ευρωκοινοβούλιο και ότι από κοινού θα μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο για την καλύτερη δυνατή χρήση και ανάπτυξη του οργανισμού. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι και τώρα στρέφομαι σε εσά. Έχετε ο καθένας το λόγο για μάξιμουμ δύο λεπτά πρώτη στον καταλογό μου είναι η κυρία Καρβάλιο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα, κυρία Λεπασάρ, να σας συγχαρώ για τον διορισμό σας. Έχετε αναλάβει δύσκολη δουλειά, ο ίδιος αναφέρατε κάποιες από τις δυσκολίες. Είναι δύσκολη δουλειά διότι είναι και πάρα πολύ σημαντική. είναι ένα θέμα υψίστης σημασίας για την Ευρώπη και μάλιστα αυξανόμενης σημασίας. Είναι τεχνικά και πολιτικά πολύ δύσκολο θέμα. Επίσης, είστε επικεφαλής ενός οργανισμού σε μια μεταβατική ε, φάση. Έχετε δυσκολίες όσον αφορά τον προϋπολογισμό, όσον αφορά την προσέλκυση του κατάλληλου προσωπικού ε, όσον αφορά τη, τα δύο γραφεία. Η ερώτησή μου είναι πώς θα λύσετε αυτά τα πρακτικά προβλήματα και τι μπορείτε να μας πείτε για να μας διαβεβαιώσετε ότι μπορούμε να βασιστούμε σε εσά. και ότι είστε σε θέση να λύσετε αυτά τα δύσκολα προβλήματα όσον αφορά δηλαδή την ε, οικονομική διακυβέρνηση, τα πολιτικά προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό ελληνικό επίπεδο, όσον αφορά τις διεθνείς ε, σχέσεις πώς μπορεί η εμπειρία σας, η επαγγελματική σας εμπειρία, αυτά που αναγράφονται στο βιογραφικό σας, θα σας βοηθήσουν ώστε να διασφαλίσετε την ομαλή ε, λειτουργία σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ κύριε Καμιλάν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Γιώχαλε Λεπασάρ, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα και θα ήθελα να σας συγχαρώ για το διορισμό σας. Με μεγάλη χαρά άκουσα τα όσα μας είπατε και ιδιαίτερα τα πολύ συγκεκριμένα σχέδιά σας όσον αφορά την εφαρμογή του νομικού πλαισίου, την, ε, δημιουργία, την ε, εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης ε, εμπιστοσύνης, Όλα τα θέματα που αναφέρατε είναι υψής της σημασίας ως Εστονή, αλλά ακόμη περισσότερο ως πρώην πρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, για την ε, Σταθερότητα στον Κυβερνοχώρο. Έχω δει την σταδιοδρομία σας τα τελευταία πέντε χρόνια. Γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα είσαστε εξαιρετικός εκτελεστικός διευθυντής του ΕΝΙΖΑ. Και γιατί τα λέω αυτά, διότι σας έχω δει εν ενεργεία, γνωρίζω πόσο καλά γνωρίζετε τα θέματα κυβερνοασφάλειας και γνωρίζω και πόσο είχατε συμμετάσχει στην προηγούμενη ε, διαδικασία κατάρτισης της νομοθεσίας. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι η κύβερνοασφάλεια δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικά των κρατών μελών. Ε, χρειαζόμαστε συμμετοχή, χρειαζόμαστε μια προσέγγιση που να διασφαλίζει την συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων ε, και επίσης θα πρέπει να συνεργαστούμε με ε, επιχειρήσεις, με πανεπιστήμια, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Εσείς πώς βλέπετε να διαμορφώνετε αυτού του τύπου η συνεργασία. Ευχαριστώ κυρία Κάμον. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια γενική θεωρητική ερώτηση και κατόπιν δύο πολύ συγκεκριμένες. Η πιο γενική μου ερώτηση είναι... Πώς ε, βλέπετε την αμυντική πολιτική στο πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας. Πιστεύετε ότι Καλά θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει περαιτέρω στην κυβερνοασφάλεια όσον αφορά την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Γενικά. Και έχω δύο πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πού θα χαράξετε τη διαχωριστική γραμμή, πώς βλέπετε τη συνεργασία ανάμεσα στον ΕΝΙΖΑ και το Κέντρο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας, το οποίο διασφαλίζει η προώθηση της έρευνας. Εσείς πώς βλέπετε τη συνεργασία, όχι μόνο ανάμεσα στο Κέντρο ε, Δεξιοτήτων, ε, αλλά και με τα εθνικά δίκτυα είναι συμπληρωματικά και ποιος θα είναι ο ρόλος του δικού σας οργανισμού όσον αφορά ε, την επιλογή των προγραμμάτων που θα ε, χρηματοδοτηθούν μέσω της ψηφιακής Ευρώπης ε, και των ψηφιακών δικτύων για την κυβερνοασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν βλέπω πουθενά τον κύριο Νινίστο, τον αντικαθιστά κάποιος. Δεν βλέπω μέχρι εκεί κάτω. Παρακαλώ, πείτε μου το όνομά σας. Yeah, uh, uh, ευχαριστώ που έχουμε τη δυνατότητα αυτή να συνομιλήσουμε μαζί σας, κύριε Λεπασάρ. Έχω μία ερώτηση. Διάβασα το βιογραφικό σας. Έχετε σπούδαση ε, εσωτερική αρχιτεκτονική ε, και αυτό ίσως μας εκπλήσει ε, εφόσον είσαστε ο κορυφαίος Ευρωπαίος για θέματα κυβερνοασφάλειας. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία ευκαιρία να πείσετε τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε ότι είσαστε το κατάλληλο άτομο για τη θέση αυτή. Στο μέλλον θα πρέπει να υποβάλλετε στρατηγικά έγγραφα σχετικά με τους ε, δείκτες απόδοσης με βάση τους οποίους θα μετράτε την ε, απόδοση του οργανισμού σας. Επίσης, το 2017 ε, είχαμε ε, θέματα ανασφάλειας ε, δικτύου στην Εστονία. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό και να μας πείτε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για ασφάλεια στα κυβερνοσυστήματά μας. Ευχαριστώ κύριε Πόρκια. Δύο λεπτά παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Εγώ έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, ήθελα να καταλάβω ποια είναι τα μέτρα που θα εφαρμόσει η ΕΝΙΖΑ για να βελτιώσει την ε, ανθεκτικότητα του δικτύου και να περιορίσει τους κινδύνους ασφάλειας όσον αφορά την εφαρμογή του 5G. Δεύτερον, ε, λέτε ότι για να αποφύγουμε μία έντονη εξάρτηση από μόνο έναν πάροχο ε, ε, ε, δικτύου θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την διαλειτουργικότητα των ε, ε, υποδομών ώστε να αποφύγουμε δηλαδή τον αποκλεισμό της χρήσης ενός μόνο παρόχου. Θα ήθελα να ρωτήσω τέλος αν υπάρχει μια στρατηγική που να έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά στη μείωση στη ρίζα της, εξάρτησης, της τεχνολογικής εξάρτησης από τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Στοσανόφσκι, θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα καταρχάς, ε, κύριε Λαπασάρ, να σας ε, συγχαρώ για τον διορισμό σας στην πολύ σημαντική αυτή θέση στον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό, του οποίου η σημασία θα αυξηθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της κυβερνοασφάλειας, γιατί έχει γίνει συζήτηση σχετικά με το αν η πιστοποίηση κάποιων προϊόντων και υπηρεσιών θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική ή να παραμείνει ε, προαιρετική. Υπό το φως της συζήτησης ε, για το δίκτυο 5ης γενιάς 5G, ε, πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχουμε υποχρεωτική πιστοποίηση διότι κάτι τέτοιο έχει και οικονομικές συνέπειες. Και από την συζήτηση δεν πιστήκαμε απόλυτα για το πού θα πρέπει να τεθεί η διαχωριστική γραμμή. Δεύτερη μου ερώτηση. Στην Επιτροπή Ήτρε πάντα τόνιζα πόσο σημαντικό είναι όλοι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί να συνεργάζονται μεταξύ τους, διότι ένας ε, απομονωμένος ευρωπαϊκός οργανισμός ποτέ δεν θα μπορέσει να διασφαλίσει απόλυτα την κυβερνοασφάλεια. Πώς βλέπετε λοιπόν το θέμα της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ασφαλείας. Εσείς, με βάση την πείρα σας, πώς θα βλέπατε τέτοια συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στους λοιπούς ευρωβουλευτές της Επιτροπής μας. Δύο λεπτά ο καθένας. Η κυρία Νίμπλερ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για τον διορισμό σας στη θέση του Διευθυντή του ΕΝΙΖΑ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο σας. Έχω μια παρατήρηση και δύο ερωτήσεις. Το Κοινοβούλιο γνωρίζετε ότι έχει αγωνιστεί για μια πολύ ισχυρή θέση του ΕΝΙΖΑ και απέναντι στα ευρωπαϊκά κρατη κράτη-μέλη και το, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ήθελα να σας καλέσω τη, το δυναμικό που σας ε, έχουμε διαθέσει να το χρησιμοποιήσετε για να ε, πληρώσετε τις ε, υποχρεώσεις σας και να ασκήσετε το έργο σας. Αυτή λοιπόν είναι η έκκλησή μου. Ο ΕΝΙΖΑ να μην είναι απλά μια γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των κρατών μελών, να είναι ένας αυτόνομος οργανισμός. Όσον αφορά, όσον αφορά το θέμα της κυβερνοασφάλειας, ο κύριος Στοσανόφσκι έθεσε μια ερώτηση της οποίας να απάντηση θα ήθελα και εγώ να ακούσω. Επίσης, όσον αφορά το τρέχον πρόγραμμα εργασιών, Πόσο έχετε προχωρήσει στη διαμόρφωσή του. Στην πράξη για την κυβερνοασφάλεια έχουμε προβλέψει και τη δημιουργία μιας ομάδας πιστοποίησης από ενδιαφερόμενους κύκλους. Πώς το βλέπετε αυτό, πού βρίσκεστε στο σημείο αυτό και τέλος έχετε πολλά καθήκοντα ποιες είναι οι βασικές σας προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες. Και αυτό θα ήθελα να μάθω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λέιτο Μαρκές, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, σας συγχαίρω για τον διορισμό σας. Η κυβερνοασφάλεια είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δεν είναι καθαρά τεχνικό, είναι και πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα διότι με την κυβερνοασφάλεια βελτιώνουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας στην ε, ε, ψηφιακή ενιαία αγορά. Δύο ερωτήσεις συγκεκριμένε και θα μιλήσω πορτογαλικά. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με τη δημιουργία του κέντρου εξειδίκευσης για θέματα κυβερνοασφάλειας. Υπάρχει ο κίνδυνος επικάλυψης αρμοδιοτήτων τώρα που έχουμε την ενισχυμένη ενίζα. Δεύτερη μου ερώτηση έχει να κάνει με την κυβερνοασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές. Υπάρχει μια εξαιρετική έκθεση του 2011 που πρέπει να ενημερωθεί ε, και χρειάζεται να εγγυηθούμε περισσότερη ασφάλεια στον τομέα αυτό που είναι τόσο σημαντικός για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ήθελα να γνωρίζω εάν έχετε κάποια ιδέα ε, για το τι θα κάνετε σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Ντελκαστήγιο. Σας ευχαριστώ για το διορισμό σας. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ και μαζί σας στην προηγούμενη ε, θητεία ε, υπό την προηγούμενη σας ιδιότητα. Μια από τις πτυχές ε, που αναφέρατε επενελειμμένα είναι η συνεργασία με τα κράτη-μέλη και ε, τους κρατικούς ε, αρμόδιους οργανισμούς, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται να συνεργαστούμε, να έχουμε μια πραγματική διεθνή πολιτική στον τομέα αυτό. Η κυβερνό ασφάλεια δεν μπορεί να είναι μόνο δική μας ε, ε, υπόθεση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε συμβατές πολιτικές με τους διεθνούς μας, διεθνείς μας εταίρους, συνεργασία ας πούμε στην διερεύνηση κυβερνο, διεθνών κυβερνοασφάλων, δημιουργία ε, διεθνούς διεθνούς συνεργασίας ε, για την δημιουργία ειδικοτήτων και δυνατοτήτων. Ε, θα ήθελα να έχω μερικές περισσότερες πληροφορίες για αυτό το τομέα της διεθνούς συνεργασίας από πλευρά σας. Ευχαριστώ και πάλι και σας συγχαίρω ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ. Κύριο Σιγκάλ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ. Έχω κάποιες... Είχα κάποιες ερωτήσεις ε, συγκεκριμένες που έθεσαν ε, άλλοι συνάδελφοι. Γι' αυτό εγώ θα περάσω στην άλλη με ερώτηση που έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό. Υπάρχει μια συμφωνία ενίζα Ελλάδος και θα ήθελα να γνωρίζω εάν τα διοικητικά προβλήματα που ε, είχαμε στο παρελθόν έχουν λυθεί. Έχουν λυθεί. Η ήταν ε, επίσημη έδρα το Ηράκλειο, ήταν πάντα δύσκολο να προσελκύσουμε εκεί προσωπικό, υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά ε, το Διεθνές ε, Σχολείο και έτσι είχαμε την περίεργη θέση να έχουμε επίσημη έδρα το Ηράκλειο, αλλά η περισσότερη δουλειά να γίνεται από την Αθήνα ένας οργανισμός με ε, de facto δύο έδρες ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ε, αν με τη νέα συμφωνία έχουν λυθεί τα βασικά προβλήματα κατά τη γνώμη σας. Σας ευχαριστώ. Thank you. Uh, ευχαριστώ κυρία Κίτενταλ ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και θα ήθελα να σας συγχαρώ για τον διορισμό σας. Έχω μία ερώτηση, διότι ε, είναι ξεκάθαρο ότι ε, έχουμε δει μόλις την αρχή των κυβερνοεπιθέσεων εις βάρος της κοινωνίας μας ε, που απειλούν τα δημοκρατικά θεσμικά μας όργανα. Γίνεται ένα και πιο δύσκολο τοπίο και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γιάννης και επανειλημμένα έχει πει ότι ε, ο κυβερνοχώρος είναι ένας χώρος όπου ε, το ΝΑΤΟ θα ε, αμήνεται εξίσου αποτελεσματικά με την άμυνα στη γη, στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Και υπάρχει άλλωστε και το άρθρο 5. Εσείς πώς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κινηθεί στο πλαίσιο αυτό, στο τοπίο αυτό με διάφορους φορείς ε, και παράγοντες, ε, διατηρώντας όμως και την κυριαρχία των κρατών μελών όσον αφορά το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κονζάλης Κασάρας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Λεπασάρα, σας συγχαίρω που διοριστήκατε εκτελεστικό διευθυντή μια πολύ σημαντική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ενισχύθηκε μετά την τελευταία ε, ε, μεταρρύθμιση και εδώ μάλιστα ζητήσαμε ε, περισσότερου πόρου για σας. Ξέρουμε ότι έχουμε μεγάλε απλέ να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια κατά τη διάρκεια προεκλογικών εξατιών σε συνιστώσει που αποτελούν την ραχοκοκαλιά του 5G και μάλιστα τον Ιούνιο, Ιούλιο συγγνώμη, έκανα μία ερώτηση όσον αφορά τον κανονισμό 534 ε, και όσον αφορά τις υποδομές 5G ε, που έπρεπε να έχει φτιαχτεί και να έχουν απαντήσει τα κράτη-μέλη μέχρι τις 30 Ιουνίου. Όμως υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν έχουν ολοκληρώσει την εργασία αυτή. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, ποιες θα είναι οι προσπάθειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε όλες, όλα τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν σε αυτό το στόχο. Διότι έχουμε μέχρι τις 30 Οκτωβρίου σύμφωνα με το τι έχω καταλάβει και σύμφωνα με το τι ισχύει για να ολοκληρώσουμε την εξολόγηση των κινδύνων. Και έπειτα θα ήθελα να γνωρίζω ποιες είναι οι, οι απόψεις σας όσον αφορά τις αμφιβολίες που υπάρχουν για τις κινέζικες ε, ε, ε, εταιρείε. Πρέπει να ανησυχούμε για αυτές τις εταιρείε από ό,τι έχω καταλάβει ή όχι. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει να πάρει το λόγο. Θα κάνω κι εγώ ένα ερώτημα γιατί μιλούσαμε για την τεχνολογία 5G σήμερα το πρωί και για να πατήσω πάνω σε ένα ερώτημα που έκανε ένας από τους συναδέλφους πιστεύετε ότι η ΕΝΙΣΑ θα πρέπει να έχει λόγο σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι χειριστές τι εννοώ, να τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου δίκτυα διαλειτουργικά, αλληλοδραστικά. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο, εχθές παρατηρήσαμε μία συμφωνία μεταξύ της Πολωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για την τεχνολογία 5G, υπογράφηκε μόλις εχθές και αναφέρεται στην ασφάλεια του δικτύου 5G και αναρωτιόμουν, θα μπορούσε η Ενίσα να προτείνει, να προωθήσει μια ενιαία, ένα ενιαίο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση από όλα τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια και την τεχνολογία 5G. Ή θα πρέπει ο καθένας, ε, το κάθε κράτος μέλος να, να υπογράφει μια ξεχωριστή συμφωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Σειρά σας τώρα, πολλές ερωτήσεις, ε, πολλές σελίδες και πραγματικά ανυπομονούμε να ακούσουμε την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε όλοι για την κυβερνοασφάλεια και για την ενίσα. Από ό,τι καταλαβαίνω από την ε, γενική κατεύθυνση των ερωτήσεων, όλοι συμφωνούμε ότι η κυβερνοασφάλεια είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό και θα πρέπει να είναι ενδελεχής η δουλειά μας. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Ήτρε για το χρόνο που έχει επενδύσει και για το ότι θεωρεί την ΕΝΙΣΑ ως ευκαιρία για ολόκληρη την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει τα ζητήματα αυτά. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα ένα προς ένα ή να τα ομαδοποιήσω κάπως γιατί έχω υπόψη μου ότι έχουμε μόνο μία ώρα στη διάθεσή μας. Θα χαρώ όμως να επιστρέψω οποιοδήποτε από αυτά τα ερωτήματα με μία επόμενη επίσκεψη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις ικανότητες μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα να σας πω ότι το όραμα που έχω για την Ενίσα όταν αποφάσισα να είμαι υποψήφιος για τη θέση αυτή το έκανα με βάση την, την ιδέα ότι οι ικανότητες μου θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες όχι μόνο για την Ενίσα αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια τα πέρασα στην ΑΝΣΥΠ, uh, uh, Δουλεύοντας με τον Αντιπρόεδρο ΑΝΣΥΠ. Κάτι το οποίο μου έδωσε μια βαθύτερη κατανόηση όχι μόνο τους εσωτερικούς μηχανισμούς της Επιτροπής και τα διαφορετικά τμήματα και τις ε, διαφορετικές ε, ε, διαφορετικά συστήματα διαμόρφωσης πολιτικής, αλλά και τα διαφορετικά κράτη-μέλη και τα εμπλεκόμενα μέρη. Παρόλα αυτά όμως μου έδωσε και τη δυνατότητα να ηγηθώ της πράξεις της κυβερνοασφάλειας που είναι και η βάση της δράσης της ΕΝΙΣΑ. Ε, κατά τη διάρκεια της, της προϋπηρεσίας μου το 2007 ήμουν αντιπρόεδρος και στη συνέχεια υπήρξα σύμβουλος για το πώς θα μπορούσε να ανταποκριθεί καλύτερα σε κυβερνοεπιθέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμουν, ίσως, ήμουν ίσως ένας από τους πρώτους ε, εθνικούς ε, εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που σκέφτηκε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια καθολική απάντηση στις ε, κυβερνοαπειλές. Επομένως, ξεκίνησα την, την, τις σπουδέ μου στην εσωτερική διακοπή κόσμηση, αλλά στη συνέχεια πέρασα έξι χρόνια να μελετώ τις ε, ευρωπαϊκές πολιτικές. Είμαι ένα άτομο που, είναι, που ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και ιδίως στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας και της κυβερνοασφάλειας, γιατί πιστεύω ότι η Ευρώπη στο σύνολό της μπορεί να κάνει διαφορά ως, τη διαφορά ως σύνολο, όχι ως μεμονωμένα μέλη. Σε ό,τι αφορά την ενίσα τώρα, ε, πιστεύω είναι σημαντικό να καταλάβει κανείς πόσο σημαντική είναι η κυβερνοασφάλεια, ποιες είναι οι τεχνικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά και πέρα από την κυβερνοασφάλεια, Υπάρχει ένα ζήτημα που διαπερνά όλα τα επίπεδα πολιτικής και ένα από τα μαθήματα που έχω, που έχω α, λάβει τα τελευταία χρόνια στην προϋπηρεσία μου είναι ακριβώς πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο κοινό παρονομαστής και πώς θα μπορούσε η ΕΝΗΣΑ να βοηθήσει στην εφαρμογή ενός κανονιστικού πλαισίου. Πιστεύω ότι βάσει του background μου θα μπορούσα να βοηθήσω στον τομέα αυτό. Θα έλεγα επίσης ότι έχω και ένα χάρισμα στο να, να καταφέρνω να συνδυάζω ε, αποτελεσματικά διαφορετικούς τομείς, ούτω ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή κυβερνοασφάλεια. Επομένως, αυτή είναι ίσως μια μικρή εισαγωγή της εμπειρίας που έχω και των ε, δεξιοτήτων μου. Αν θυμάμαι καλά, το ζήτημα του κατά πώς βλέπω εγώ τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη και πώς μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτά τα οποία κάνει η ΕΝΙΣΑ. Η ΕΝΙΣΑ έχει διαφορετικές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά εμπλεκόμενα μέρη, αφενός ως συμβουλευτικό σώμα και αφετέρου σε ό,τι αφορά την πράξη κυβερνοασφάλειας. Πιστεύω ότι και η κυρία Νίμπλερ έκανε την ίδια ερώτηση. Από όσο ξέρω εγώ, έχει υπάρξει μια πρώτη έκκληση, προς ανταπόκριση, μια πρώτη πρόσκληση, ούτω ώστε τα εμπλεκόμενα μέρη που θα ήθελαν να συμπεριληφθούν στις διαδικασίε αυτές να κάνουν αιτήσει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Η ΕΝΙΖΑ είναι μια ομάδα που αποτελείται από διάφορες υποομάδες ε, διαφορετικών ενδιαφερόντων και θα πρέπει να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της, της κοινωνίας αλλά και διαφορετικών τμήματων της κοινωνίας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την ακαδημία, θα πρέπει να κοιτάξουμε τις καταναλωτές, θα πρέπει να κοιτάξουμε την ερευνητική κοινότητα. Και η Ενίζα θα πρέπει να έχει πλήρη συνείδηση του ότι πόσο ευρεία θα πρέπει να είναι η δράση της και πόσο θα πρέπει να καλύπτει όλα τα διαφορετικά, όλους τους διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας. Νομίζω υπήρξε και ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά uh, τον οδικό χάρτη. Πιστεύω ότι αν κοιτάξουμε τη δομή του προγράμματος αυτού, υπάρχουν έξι προτεραιότητες, οι οποίες το πρόγραμμα εργασίας, η δομή είναι καλή και μπορεί να λειτουργήσει για το καινούριο κανονιστικό πλαίσιο. Αν κοιτάξουμε όμως, αν εξετάσουμε τους στόχους που πρέπει να φτάσουμε, ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς της ΕΝΙΣΑ είναι να μπορεί να παρέχει έρευνες, να μπορεί να διοργανώνει events για να έρθουν τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη σε επαφή. Κάτι το οποίο, στο οποίο θέλουμε να δώσουμε έμφαση είναι να μπορέσουμε να χτίσουμε δίκτυα εμπειρογνωμόνων σε διαφορετικούς τομείς, ούτω ώστε να έχουμε μια βάση δεξιοτήτων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, που να μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να μπορούμε να, παρέχουμε βοήθεια, αλλά και να, να χτίσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Και αυτό μπορεί να γίνει σε πολύ συγκεκριμένους ε, τομείς αυτό που εξετάζουμε δεν είναι μόνο το πώς μπορούμε να συντονίσουμε, ή πώς να επικοινωνήσουμε τις διάφορες μελέτες, αλλά και πώς να ε, συνοδεύσουμε όλες αυτές τις δημοσιεύσεις με την ανάλογη ανάπτυξη των δικτύων ε, εμπειρογνωμόνων. Οι δεξιότητες αυτές και οι εμπειρογνώμονες αυτοί δεν ε, προέρχονται αποκλειστικά από το δημόσιο τομέα, προέρχονται και από τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί η Ευρώπη ε, είναι πλούσια σε, σε γνώση ασφάλειας. Πρέπει να βρούμε τρόπο λοιπόν πώς να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη γνώση αυτή και πώς μπορεί η Ένωση να αξιοποιήσει όλα αυτά τα δίκτυα. Υπήρξε και ένα ερώτημα για τις αρμοδιότητες της ε, κυβερνοασφάλειας τη πράξεις κυβερνοασφάλεια Θα είναι συμπληρωματική τη ΕΝΙΣΑ. Όπως ανέφερα προηγουμένως, ένα από του ένας από τους της ΕΝΙΣΑ είναι να μπορεί να προσφέρει έρευνες και μελέτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει και με διαφορετικούς κινδύνους που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας με ενδεχόμενες μελλοντικέ απειλές. Αυτό η ΕΝΗΣΑ το κάνει σε συνεργασία με, πολλά άλλα οργανι... με πολλούς άλλους οργανισμούς και Ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί, ακόμη περισσότεροι, που θα μπορούσε να συνεργαστεί από κοντά η ΕΝΗΣΑ, ούτως ώστε να πολλαπλασιάσει τη γνώση της, να βελτιώσει το δίκτυο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, για παράδειγμα, πώς λειτουργεί η κυβερνοασφάλεια στην ενέργεια, πώς λειτουργεί η κυβερνοασφάλεια στις μετακινήσεις ή στα προϊόντα καθημερινής χρήσης. Υπάρχουν οργανισμοί που γνωρίζουν τον κάθε διαφορετικό τομέα και αυτό είναι κάτι που η ΕΝΙΣΑ θα μπορούσε να το ακτινοποιήσει. Σε ό,τι αφορά το μέλλον, το δίκτυο δεξιοτήτων της ΕΝΙΣΑ θα μπορούσε να αξιοποιήσει κάποιες από αυτές τις νέες τεχνολογίες αλλά και κάποιες από τις προκλήσεις, διαδικαστικές προκλήσεις που έχουν ε, προκληθεί από όλες αυτές τις τεχνολογικές πρόοδους. Αυτή είναι τομείς που η ΕΝΙΣΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της. Έχει ανάγκη την ερευνητική κοινότητα, έχει ανάγκη την βιομηχανία για να μπορέσει να καταλάβει ποιες είναι οι δυνατότητες και ποιοι είναι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Και μετά μπορούμε να πούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να υπερκάμψουμε κάποια εμπόδια, κάποιες προκλήσεις. Έτσι λοιπόν η, η σύσταση ενός τέτοιου δικτύου είναι πολύτιμη αν καταφέρουμε να το χτίσουμε, θα είναι ένας πραγματικά αξιόλογος σύμμαχος στην δουλειά της ΕΝΙΣΑ. Τώρα, μέσω της δουλειά της ως κέντρο εμπειρογνωμόνων η ΕΝΙΣΑ ε, διαθέτει ένα πλούτο α, πληροφοριών. Έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα χάρτη λήψεων, αν θέλετε, που θα μπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θα πρέπει να λειτουργήσουμε γρήγορα, να αντιδράσουμε γρήγορα. Υπήρχε ένα ερώτημα για το συμβάν στην Εστονία, το ID Chip συμβάν στην Εστονία το 2017. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα για γιατί χρειαζόμαστε ε, μία αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το συγκεκριμένο chip είχε πιστοποιηθεί από κάποια εργαστήρια. Όταν ε, εντοπίστηκε το πρόβλημα, το εργοστάσιο που είχε χορηγήσει το πιστοποιητικό δεν είχε λειτουργήσει υπό έγκριση. Αυτό που χρειαζόμαστε όμως και ποιο είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια, είναι κάτι το οποίο δεν θα επιτρέπει, για παράδειγμα, το ενδεχόμενο οι Πορτογάλοι να μην εμπιστεύονται ένα πιστοποιητικό που έχει χορηγηθεί από το χύψη εργαστήριο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό πιστοποιητικό το οποίο να το εμπιστεύονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αν έχουμε εθνικά πιστοποιητικά τότε δεν θα είναι αξιόπιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούμε να επωφεληθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο από τα πιστοποιητικά αυτά. Το να δημιουργούμε εμπιστοσύνη και διαφάνεια, κάτι το οποίο ε, είναι κάτι που θα συνοδεύει το πιστοποιητικό, είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα τώρα για την τεχνολογία 5G, υπήρχαν αρκετά ερωτήματα για την τεχνολογία 5G. Επιτρέψτε μου να τις ομαδοποιήσω λίγο όλες αυτές τις ερωτήσεις και ελπίζω να απαντήσω σε όλες. Το ζήτημα... Τώρα βρισκόμαστε εν μέσω της διαδικασίας εξέτασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια σύσταση για την Άνοιξη Υπάρχουν κάποια πρώτα κράτη-μέλη που κάνουν εκτιμήσεις και μελέτες κινδύνου. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι από όσο ξέρω. Υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν έχουν συνεισφέρει, δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που να έχουν συνεισφέρει, αλλά ίσως να, να είμαι λάθος, ε, θα μπορούσατε να το ελέγξετε καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σημείο αυτό. Η δεύτερη φάση τώρα έχει να κάνει με την συλλογή των στοιχείων και την εκπόνηση μιας μελέτης κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΝΙΣΑ, το ξέρω ήδη γιατί είχα κάποιες επαφές με συναδέλφους στην ενίσα που με υποδέχτηκαν και με ενημέρωσαν τους ώστε να είμαι καλά ενημερωμένος πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου. Η Ενίσα έχει κάνει μια συγκεκριμένη ανάλυση απειλών σε σχέση με την τεχνολογία 5G. Πιστεύω ότι η Ενίσα είναι ένας εξαιρετικός φορέας για να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε τις τεχνικές γνώσεις που χρειάζονται. Αυτό που μπορώ να σας πω βεβαίως είναι ότι αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο ζήτημα. Όταν αναφερόμαστε στην τεχνολογία 5G δεν είναι κάτι που μπορούμε απλά να τσεκάρουμε ένα κουτί και να πούμε ε, τι μπορεί να γίνει. Θα πρέπει η τεχνολογία 5G να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι των ερευνών που κάνουμε διαρκώς. Υπήρξε το ερώτημα ποια θα, θα πρέπει να είναι η προσέγγιση των κρατών μελών. Και η, πρόδρο και η πρόεδρος με ρώτησε αν θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο. Πιστεύω ότι η σύσταση της Επιτροπής κατά κάποιο λόγο ήδη προτείνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, μια συνεργασία μαζί με τα κράτη-μέλη βεβαίως, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια μελέτη εκτίμησης κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μετά μπορούμε να αποφασίσουμε αν χρειαζόμαστε κοινή δράση, αν χρειαζόμαστε κοινά μέτρα, τόσο ώστε να αντιμετωπίσουμε κάποιους από αυτούς τους κινδύνους. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δουλειά της ΕΝΙΖΑ να πει αν θα πρέπει να κάνετε αυτό ή το άλλο. Η ΕΝΙΖΑ αυτό που μπορεί να κάνει είναι να προσφέρει τεχνογνωσία και γιατί τα δεδομένα δεν έχουν συλλεχθεί ακόμα, δεν μπορώ να το, να το προκρίνω και να σας πω τι προτείνει η Ενίσα; ή κατά πόσο το επίπεδο του κινδύνου είναι υψηλό ή χαμηλό. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι η ενισα ετοιμάζει την μελέτη αυτή και θα την παρουσιάσει στην Επιτροπή. Νομίζω ότι το, όριο, το χρονικό όριο ήταν ο Σεπτέμβριος. Θα χαρώ όμως να σας πω περισσότερα και να, και να επιστρέψω όταν θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή. Ελπίζω να έχω ακόμα χρόνο. Ρωτήσατε αν η πιστοποίηση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Το παρόν πλαίσιο είναι ε, προαιρετικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν το αποφασίσει ο νομοθέτης ε, δεν ε, θα μπορέσουν να εισαχθούν κάποια στοιχεία στο νομοθετικό πλαίσιο. Πρόκειται για πολιτική απόφαση και ε, γνωρίζετε καλά το θέμα από τις διαπραγματεύσεις για την πράξη για την κυβερνοασφάλεια. Επελέγει τότε να διατηρηθεί προαιρετική η πιστοποίηση. Ο Ενίζα πολύ ευχαρίστως θα συμβάλλει στον διάλογο ε, σχετικά με το ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή ενεργούμε με βάση την πράξη για την κυβερνοασφάλεια που έχει υιοθετηθεί και που προβλέπει προαιρετικό πλαίσιο. Τέθηκε ερώτηση σχετικά με τη συνεργασία του ΕΝΙΖΑ με διάφορους οργανισμούς. Ήδη αναφέρθηκα εν μέρη σε αυτό η συνεργασία αυτή ε, γίνεται προς δύο κατευθύνσεις. Ο Ενίζα ήδη έχει μνημόνια κατανόησης ε, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, ε, την Europol και άλλους ώστε ο ΕΝΙΖΑ να μπορεί να τους υποστηρίζει και στις δικές τους εργασίες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι σχέσεις αυτές. Αναφέρθηκα στην ιδέα δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου εμπειρογνωμόνων ε, και να έχουμε μια δεξαμενή ικανοτήτων. Αυτό απαιτεί προσωπικό και πόρους από τους διάφορους οργανισμούς και ε, σκοπεύω να συνομιλήσω με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανισμών και ε, μία εβδομάδα μετά την πιθανή ανάληψη των καθηκόντων μου θα γίνει μια συνάντηση, αλλά και με άλλους ε, οργανισμούς όπως είναι ο ΕΑΖΑ και λοιπά θα ε, ήθελα να συνεργαστώ περισσότερο ε, διότι και εκείνοι μπορούν να επεφεληθούν από τη δουλειά της ΕΝΙΣΑ αλλά και εκείνοι μπορούν να μας υποστηρίξουν στις δικές μας εργασίες. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η καθηγήτρια Νίμπλερ ρώτησε σχετικά με την θέση του ΕΝΙΖΑ. Όχι, δεν είναι γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε είναι το κατοικίδιο, το σκυλάκι κάποιου κράτους μέλους. Ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στον χώρο της κυβερνοασφάλειας μία από τις λέξεις κλειδιά είναι η αλληλεξάρτηση. Τα κράτη-μέλη εξαρτώνται το ένα από το άλλο, ε, εξαρτώνται από την δυνατότητα ο ένας του άλλου ε, να αντιδρούν σε κυβερνοεπιθέσεις. Δεν είναι ανεξάρτητα λοιπόν με αυτή την έννοια και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να ε, οικοδομήσουμε τις σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες. Από την άλλη, οι συμβουλές και η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΝΙΖΑ δεν ε, μπορούν να καπηλευθούν από μία ομάδα ενδιαφερομένων και... Μάλλον ε, αυτό είχε κατά νου όταν είπε ότι ο ΕΝΙΖΑ θα πρέπει να είναι ένας ανεξάρτητος, ένας αυτόνομος ευρωπαϊκός οργανισμός. Όσον αφορά το τρέχον πρόγραμμα εργασίας, κάτι που θα ήθελα να δω εγώ θα ήταν ε, τα αποτελέσματα των εργασιών μας να μην είναι μόνο εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις, αλλά να δούμε και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων, ε, μια δεξαμενή ικανοτήτων ε, και πώς μπορούν αυτά να ε, υποστήριξουν τις εργασίες του ΕΝΙΖΑ. Νομίζω ότι επίσης απάντησα ε, όσον αφορά την ε, ομάδα που αναφέρατε και ποιες είναι οι προτεραιότητες κλειδιά μας για τους επόμενους μήνες. Η ημέρα που πιθανότατα να αναλάβω τα καθήκοντά μου είναι και η μέρα που θα πρέπει να υιοθετηθεί το πρόγραμμα εργασίας, το πρόγραμμα εργασιών του ΕΝΙΣΑ και το πρώτο που θα πρέπει να κάνω θα πρέπει να είναι να δω τι μπορεί να κάνει ο ΕΝΙΣΑ. Έχει όλα όσα χρειάζεται για να μπορέσει να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα εργασιών. Από ό,τι γνωρίζω, το πρόγραμμα εργασιών ε, ήδη αντικατοπτρίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο, το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Και μάλιστα περιλαμβάνει συγκεκριμένη δράση ε, σχετικά με ανανέωση της ε, μελέτης. Ε, ο ΕΝΙΣΑ όμως χρειάζεται να έχει και τους διάφορους πόρους για να μπορεί να εφαρμόσει το νέο πρόγραμμα εργασιών. Υπάρχει ένας νέος τομέας που είναι η πιστοποίηση κυβερνοασφάλειας και ο ΕΝΙΖΑ θα πρέπει να οικοδομήσει δυναμικό όχι μόνο όσον αφορά το προσωπικό, αλλά και όσον αφορά τις διαδικασίες, την κατανόηση, τη γνώση ε, και το δίκτυο. Ναι, ναι, θα κλείσω. Νομίζω λοιπόν ότι ε, όσον αφορά τα θέματα ουσίας, αυτά θα είναι οι πρώτες μου προτεραιότητες. Ε, ήδη ε, έχω σημειώσει αυτό που είπατε για τον προϋπολογισμό. Πρέπει να διευκολύνουμε την ε, νέα συμφωνία που υιοθετήθηκε την Άνοιξη, που προβλέπει κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, επίσης παράρτημα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. και κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει λοιπόν να κλείσει το θέμα αυτό και θα επικοινωνήσω με τις ελληνικές αρχές για να μπορέσω ε, να διευκολύνω και να επιταχύνω τη διαδικασία επικύρωσης αλλά και την εφαρμογή της νέας συμφωνίας. Ο οργανισμός χρειάζεται βεβαιότητα σχετικά με το νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο εργαζόμαστε και εν θα πρέπει να... Μέρος αυτού είναι να εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εξαλείψουμε τις επικαλύψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ, θα πρέπει να εξαλειφθούν. Ε, και είναι κάτι που θεωρώ προτεραιότητα. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στις δεξιότητες, ε, τις προσλήψεις. Χρειαζόμαστε ικανούς ανθρώπους ε, και σκοπεύω να φροντίσω ο Ενίσα να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αναφέραμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. So Σας ευχαριστώ πολύ για την εισήγησή σας. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι που Υποβάλατε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ε, ευχόμαστε καλή επιτυχία σε εσά και στην Ενίσα. Ελπίζουμε να πάρετε και να οριστικοποιηθεί ο διορισμός σας. Ε, θα ε, πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα στην πορεία. Θέλω να σας πω ότι θα ήθελα να καλωσορίσω την Επιτροπή Ήτρε στην Ενίζα. Οποτεδήποτε έχετε ε, χρόνο, δεν ξέρω αν κάνετε τέτοιες αποστολές, επισκέψεις, αλλά θα ήταν σημαντικό να καταλάβετε πώς λειτουργεί η Ενίζα και να καταλάβετε, δείτε από κοντά ποιες είναι οι προκλήσεις. Πάντως έχετε ανοιχτή πρόσκληση από πλευράς μου, αν έχετε το χρόνο. Μάλιστα. Θα πρέπει να βρούμε χρόνο, ε, γιατί πρέπει να έρθουμε στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πολύ. Uh, we move to the next item. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Αγαπητοί συνάδελφοι, επόμενο σημείο στην ημερησία μας διάταξε είναι η ανταλλαγή απόψεων με τη Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης. Παρακαλώ, όσοι έχετε μεταξύ σας συνομιλίες να βγείτε από την αίθουσα. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Ντίτε Γιούλ Γιόγκρισεν είναι νεοδιοριστής Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σα ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα και προσβλέπουμε να ακούσουμε τα σχέδιά σας. Έχουμε, έχετε, έχετε ιδέες, θέλουμε να δούμε πώς ε, ε, βλέπετε τα πράγματα εσείς και ιδιαίτερος πιστεύω πως οι συνάδελφοι θα ήθελαν να ακούσουν περισσότερα για την κατάσταση προόδου των εθνικών προγραμμάτων ενέργειας και, ε, το, και κλίματος για την περίοδο 2021 με 2030. Έπειτα και τις επερχόμενες ε, νομοθετικές προτάσεις για την επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης. Συνάδελφοι, έχουμε νομίζω κάποιο χρόνο για όλα αυτά, ίσως μια ώρα στη διάθεσή μας. Και ε, βεβαίως ε, θα ήθελα να σας ζητήσω να ακούσετε προσεκτικά τη Γενική ε, Διευθύντρια και να τη ρωτήσετε τα όσα θα επιθυμούσατε να μάθετε σε αυτό το στάδιο από την Επιτροπή. Παρακαλώ λοιπόν κυρία Διευθύντρια έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Βαλεάν, ε, Αντιπρόεδρη, ε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές και συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να έρθω σήμερα εδώ. Σας συγχαίρω όλους για την εκλογή σας ε, στο Επιτροπή ε, και σας Πρόεδρε, καθώς και για τα νέα μέλη της, του Ευρωκοινοβουλίου. Ξέρω πως είστε αρκετοί νέοι ευρωβουλευτές. Καλωσορίσατε σε αυτή τη σημαντική ε, επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Μπορώ να πω εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα ε, εξ ονόματος του Γενικής Διεύθυνσης Συνέργειας ότι προσβλέπω σε μια στενή και επικοδομητική συνεργασία μαζί σας με βάση την πολύ καλή εμπειρία που είχαμε τα τελευταία πέντε ε, χρόνια. Όπως είπατε, μόλις ανέλαβα τη θέση μου ως Γενική Διευθύντρια ε, της Διεύθυνσης Ενέργειας, ε, ξεκίνησα την 1η Αυγούστου, αλλά όπως ήταν ήσυχος μήνας και έτσι είχα το χρόνο να τακτοποιηθώ στο γραφείο μου. Επειδή μόλις ξεκίνησα, θα ήθελα να αποτίσω φόρο το ημίς στον προκάτοχό μου, Ντομινίκ Στουρί, που γνωρίζετε καλά όσοι βρισκόσασταν σε αυτή την Επιτροπή στην τελευταία θητεία γιατί ήταν ιδιαίτερα αφοσιωμένο ε, στη... και για τον τρόπο με τον οποίο ηγήθηκε τη Γενική Διεύθυνσης Ενέργειας τα περασμένα πέντε χρόνια και την εργαστή συνεργασία που είχατε μαζί του ε, τα τελευταία πέντε χρόνια. Για όσους δεν με γνωρίζετε, εργάζομαι εδώ και 27 χρόνια ως υπάλληλο στην Επιτροπή, περισσότερο στην, ε, πολιτική ανταγωνισμού και στην εμπορική πολιτική και τα ζητήματα ε, που αφορούσαν τον ΟΗΕ. Σε όλες αυτές τις θέσεις ασχολήθηκα με την ενεργική πολιτική με κάποιο τρόπο και γι' αυτό τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένη που έχω την ενέργεια στο επίκεντρο των όσων κάνω συνεργάζομαι μαζί εδώ σημαίνει εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος για την ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατευθυντήριες γραμμές θα μας οδηγήσουν και στις επόμενες μας κατευθυντήριες πολιτικές ε, που ορίστηκαν και από την Επίτροπο για την Πράσινη ε, Συμφωνία. Η πρώτη μου δημόσια εμφάνιση είναι σήμερα, από τότε που ανέλαβα καθήκοντα και δεν είναι σύμπτωση που επισκέπτομαι πρώτα εσάς, γιατί είστε άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης και συνομοθέτες. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι ζωτικό κομμάτι της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων της δημοκρατίας μας και βρίσκεται κοντά ε, στους Ευρωπαίους πολίτες. Όπως σας ανέφερα, τα τελευταία θητεία, τα περασμένα πέντε χρόνια. Η Επιτροπή μου, ε, η Διεύθυνσή μου και η Επιτροπή αυτή έχουν συνεργαστεί στενά και η Επιτροπή σας ήταν ε, καθοριστική σημασία για την υιοθέτηση ε, σημαντικών νομοθετικών πράξεων. Όπως είχα την δυνατότητα να συζητήσω μαζί σας, ήδη στόχος είναι να συνεχίσουμε αυτή τη στενή και παραγωγική συνεργασία τα επόμενα πέντε χρόνια. Εγώ είμαι ανοιχτή σε έναν μόνιμο διάλογο με εμένα την ίδια και το επιτελείο μου. Στην σημερινή μου δήλωση θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για το πού βρίσκεται η ενεργειακή πολιτική επί τη βάση της νομοθεσίας που έχει περάσει και να αναφερθώ στις τέσσερις εκθέσεις που ζητήσατε την τέταρτη έκθεση προόδου για την Ενεργειακή Ένωση, την έκθεση για την ανανεώσιμε ενέργειες, την πρόσφατη έκθεση τη για τι ε, ε, εθνικέ εκθέσει. Ε, εθνικά σχέδια και βεβαίως θα δεχτώ ερωτήσεις και θα πω και δύο λόγια όσο γι' αυτό γίνεται για το τι μας αναμένει τα επόμενα χρόνια. Πρώτα λοιπόν που βρισκόμαστε. Έχουμε θεσπίσει στόχους για το 2020 και έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο ολόκληρη την Ένωση για την επίτευξή τους τα τελευταία χρόνια. Αλλά όπως ίσως να έχετε δει σε κάποιες από τις εκθέσεις η πρόοδος έχει κάπως καθυστερήσει σε κάποιες ε, τομείς και γι' αυτό χρειάζεται να μπορέσουμε να συναντήσουμε, ε, να τηρήσουμε αυτούς τους στόχους που εμείς οι ίδιοι έχουμε θεσπίσει. Τώρα, ε, η γενική τάση είναι μειωτική όσον αφορά την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό που είναι ενδιαφέρον να το δούμε από ευρύτερο πλαίσιο οικονομικό και ευρωπαϊκό είναι ότι καταφέραμε να μειώσουμε τις εκπομπές ενώ έχουμε αυξήσει την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη και γι' αυτό έτσι έχουμε καταργήσει το μύθο ότι πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στην μείωση των εκπομπών και την ανάπτυξη της οικονομίας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και τα δύο, αλλά είναι σημαντικό να προσέξουμε για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και τους δύο αυτούς στόχους. Υπάρχει ενέργεια, έχει υπάρξει μια πρόοδος, αλλά έχει υπάρξει μια στασιμότητα από το 2015 και ενώ η κατανάλωση έχει αυξηθεί. Πρέπει σε αυτό να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Έχουμε επίσης ε, συγκεκριμένες task force, πρέπει αυτές να κινητοποιηθούν για να φτάσουμε τους στόχους του 2020 και βεβαίως συνεχίζουμε να εκμεταλλευόμαστε το δυναμικό που έχουμε όσον αφορά την ενεργειακή επάρκεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια, 11 κράτη-μέλη έχουν ήδη επιτύχει το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας που αντιστοιχεί στους στόχους, εθνικούς στόχους 2020. Γενικώ ε, θα επιτύχουμε το επίπεδο φιλοδοξίας, αλλά και πάλι το, ο ρυθμός έχει κάπως μειωθεί τα τελευταία χρόνια και τα κάτι μέλη θα πρέπει να επιταχύνουν μέχρι το 2020 και πέρα από αυτό για να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους. Τώρα όσον αφορά την νομοθεσία, τα περασμένα πέντε χρόνια μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε ένα εντυπωσιακό ε, φάσμα ε, ε, νομοθεσίας για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Να αναφερθώ σε ένα που είναι ακόμα εκρεμή ακόμα δηλαδή η, η ετικετοθεσία, από ό,τι κατάλαβα, θα διοριστεί νέος εισηγητής για να την καταστήσει τον προηγούμενο εισηγητή, καθώς και του σκιώδης και ελπίζουμε πως αυτό θα προχωρήσει σύντομα, ώστε να ξεκινήσουμε τους τριμερείς διαλόγους και να ολοκληρωθεί σύντομα αυτή η σημαντική νομοθεσία που θα έχει πραγματικό αντίκτυπο στον περιορισμό εκπομπών και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν μιλώ για νομοθεσία είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η νομοθεσία ε, είναι ισχυρή όταν εφαρμόζεται σωστά. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την εργασία μας ώστε αυτοί οι νομοθεσίες που έχουμε γκρίνει να εφαρμόζονται. Τα κράτη-μέλη το προσπαθούν αυτό. Και είναι πολύ σημαντική η νομοθεσία, αλλά και εξίσου σημαντική είναι η επιβολή της και η εφαρμογή της. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα κρατημέλη και να τα καθοδηγήσουμε εκεί όπου αυτό χρειάζεται για την μεταγραφή και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ένα από τα πολύ σημαντικά επιτεύγματα των περασμένων πέντε ετών είναι οι νέοι κανόνες περί διαχείρισης της ε, ενέργειας όπου κάθε κράτος υποχρεούται να υποβάλει εθνικό σχέδιο δράσης τα οποία έχουν υποβληθεί ε, πριν το τέλος του καλοκαιριού και τα τελικά σχέδια θα υποβληθούν πριν το τέλος του χρόνου. Κάθε ένα από αυτά τα σχέδια, τα εθνικά σχέδια οφείλουν να δίνουν μια συνολική εικόνα για το πώς προτίθεται να ανταποκριθεί και να επιτύχει τους στόχους ε, του 2030. Αυτό είναι βασικό στοιχείο στην εφαρμογή και παρέχει συγκρίσιμες ε, πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για, την πρώτη φορά, για πρώτη φορά στα χρονικά. Πρόκειται για ένα μέσο διαλόγου και συνεργασίας με τα κράτη-μέλη για να επιτευχθούν οι συμπεφωνημένοι στόχοι σε εθνικό επίπεδο. Είναι μια νέα έννοια για όλους. Έχουμε δημοσιεύσει την πρώτη έκθεση για τον αντίκτυπο των σχεδίων αυτών ε, πριν το καλοκαίρι, όπου δώσαμε συγκεκριμένες υποδείξεις για το πώς κάθε χώρα θα μπορούσε να βελτιώσει το σχέδιο της, ώστε να οριστικοποιηθούν τα σχέδια αυτά πριν τα τέλη του έτους. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες για κάθε ένα από αυτά τα ε, εθνικά σχέδια, αλλά μπορώ να πω το πολύ θετικό στοιχείο ότι βλέπουμε μεγάλη ε, συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία που είναι νέα και όπου βλέπουμε να υπάρχουν πολλές ε, όπου μάλλον υπάρχει πολλή διακυβερνητική συνεργασία. Βλέπουμε λοιπόν αφοσίωση, προσήλωση στο να εκπονηθούν καλά εθνικά προγράμματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έλλειψη όσον αφορά το παγκόσμιο αντίκτυπο αυτών των σχεδίων για την επίτευξη του στόχου, των στόχων του 2030 για την ανανεώσιμη ενέργεια και την επάρκεια σε ενέργεια. Δεν είναι πολύ αργά να συμπληρωθεί αυτό το κενό. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη τώρα γιατί οι κυβερνήσει έχουν μέχρι το τέλο του χρόνου να ολοκληρώσουν τα εθνικά του ε, προγράμματα. Να πω ότι αυτή η διαδικασία βασίζεται στη διαφάνεια, το διάλογο και την επικοινωνία ε, και βεβαίως το Ευρωκοινοβούλιο βοηθά στη συμμετοχή στη συζήτηση ώστε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων. Τώρα, προσβλέποντας την επόμενη ε, Επιτροπή να πω δύο λόγια. Υποψήφιο ε, ε, πρόεδρος της Επιτροπής, ε, Ούσουρα Φαντελάιεν, μίλησε για ένα φιλόδοξο πράσινο σύμφωνο, μια πράσινη συμφωνία ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί στην πράσινη παραγωγή ενέργειας μέχρι το 2050. Έχουμε ο 50% των εκπομπών που οφείλονται στην παραγωγή ενέργειας, γι' αυτό και η ενεργειακή πολιτική θα είναι πολύ σημαντική γιατί η πράσινη αυτή ε, συμφωνία ε, με βάση και τις νομοθεσίες που έχουμε θετήσει τα τελευταία πέντε χρόνια. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν είναι περιορισμένο η εργαλειοθήκη μας στην νομοθεσία. Έχουμε και διάφορες μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα συνεχίσουν να έχουν πολύ μεγάλη σημασία όσον αφορά το Green Deal, όπως ας πούμε συνεργασία για τη μετάβαση από τον άνθρακα για τις περιφέρειες που εξαρτώνται ακόμα πολύ από τον άνθρακα. Έχουμε και τη, την πρωτοβουλία για τον καθαρό ε, άνθρακα ε, και στον πολιτικό ε, άξονα είχε δεσμευθεί, έχει δεσμευθεί η Πρόεδρος να προτείνει μια πράσινη συμφωνία καθώς και ένα κλιματικό νόμο για την ουδετερότητα του κλίματος. Μίλησε για την αύξηση των στόχων περιορισμού ε, των εκπομπών μέχρι το 2030 και ε, να ηγηθεί μιας σχετικής πρωτοβουλίας. Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα ε, ε, building blocks, δηλαδή λύθη επί των οποίων να οικοδομηθεί το, ε, όπως ας πούμε το, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα, το Ευρωπαϊκό ένα επενδυτικό πρόγραμμα για το κλίμα, επενδύσεις με στρατηγική για πράσινη χρηματοδότηση, ε, και η προστασία του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Ε, σήμερα δεν μπορώ να σας πω περισσότερα για όλα αυτά, γιατί οι πολιτικές κατευθύνες γραμμές έχουν θεσπιστεί και πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε να εξετάζουμε πώς θα προχωρήσουμε. Αλλά αυτό βεβαίως θα είναι υπόθεση για την νέα ε, Επιτροπή. Δεν θα πω λοιπόν περισσότερα, αλλά πραγματικά προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας καθώς θα ε, ε, προωθήσουμε την πράσινη αυτή συμφωνία, το Green Deal και τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που ήθελα να τονίσω. Η ενεργειακή πολιτική βεβαίω ξεπερνά τα όσα εγώ σας ανέφερα σήμερα, αλλά ε, λόγω του χρόνου και λόγω του ότι θα ήθελα να ακούσω σχόλια δικά σας και ερωτήσει, θα σταματήσω σε αυτά. Ανάμεσα σε άλλα θέματα που είναι εξίσου σημαντικά με την ενεργειακή πολιτική είναι βέβαια η ασφάλεια ε, ανεφοδιασμού, το να είναι πιο προσιτή ενέργεια για τους καταναλωτές, καταπολέμηση της ε, ε, ενεργειακής φτώχειας, ε, η ενεργειακή δημοκρατία και η διεθνής επιτυχή της ενεργειακής πολιτικής. Τώρα βρισκόμαστε στα μέσα μιας ιστορικής μετάβασης, έχουμε προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και ελπίζω πως η εφαρμογή της πρόσφατης νομοθεσίας και κυρίως το πακέτο για την καθαρή ενέργεια για όλους θα ε, βοηθήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η μετάβαση μέχρι το 2024. Πιστεύω πως θα έχουμε έτσι εξασφαλίσει μια δίκαιη ε, μετάβαση. Ε, να τελειώσω λέγοντας πως βλέπω ε, το έργο μου ως Γενικής Διευθύντριας σε, σε στενή συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε δύσκολα θέματα και πολλές φιλοδοξίες. δεν θα συμφωνούμε πιθανότατα για όλες τις πτυχές, αλλά είμαι βεβαία πως θα συνεργαστούμε επικοδομητικά ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, καταρχάς που ήρθατε και για την παρουσίασή σας. Συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε συνήθως από τους συντονιστές και κατόπιν θα ακούσουμε άλλους ευρωβουλευτές που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Η κυρία Καρβαϊό, ο συνήθως σήμερα. Δύο λεπτά παρακαλώ. Please. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Γενική Διευθύντρια. Ήθελα καταρχάς να συγχαρώ εσάς, της υπηρεσίες σας, ε, τον προκατοχό σας και τον ε, Επίτροπο Καγιέτε για την εντυπωσιακή δουλειά που έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστούμε για όλη αυτή τη δουλειά. Είναι τομέα όπου έχουμε δει πραγματικά πολλά αποτελέσματα. Η ερώτησή μου συνδέεται άμεσα. Αναφέρατε το καθήκον της εφαρμογής της νομοθεσίας. Και είπατε ότι θα εφαρμοστούν όλα αυτά στα διάφορα κράτη-μέλη όπου επικρατούν διάφορες συνθήκες, στα κράτη-μέλη με όλες τις ιδιαιτερότητες. Η ερώτησή μου λοιπόν συνδέεται με κάτι που είπατε. Η κυρία Ούρσουλα Φαντερ Λάιεν ε, δήλωσε τις, ε, περιέγραψε τους φιλόδοξους στόχους της όσον αφορά το κλίμα. Πώς πιστεύετε ότι αυτά θα επηρεάσουν το νομοθετικό πακέτο που έχει ανακοινωθεί. Το σκέφτεστε αυτό, διότι άλλο το να είναι κανείς φιλόδοξος όσον αφορά τους στόχους και άλλο το να είναι ρεαλιστής σχετικά με το πώς αυτά θα εφαρμοστούν. Και η τελευταία μου ερώτηση συνδέεται ακριβώς με αυτές τις φιλοδοξίες. Ε, θέλουμε να είναι όχι απλά φιλοδοξίες, αλλά να δούμε αποτελέσματα. Και για να δούμε αποτελέσματα θα πρέπει να φροντίσετε οι κοινωνίες μας, ε, η οικονομία μας ε, να είναι σε θέση να παρουσιάσει αποτελέσματα. Και θα πρέπει επίσης να υπάρχει και η απαραίτητη τεχνολογία, την οποία δεν έχουμε ακόμα. Χρειαζόμαστε περισσότερες έρευνες, για παράδειγμα η δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα δεν ε, έχει προχωρήσει αρκετά. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε πολλά ακόμη για να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας. Σας ευχαριστώ πολύ για όλη τη δουλειά που έχετε κάνει. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ κύριε Στίκα. Παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Διευθύντρια, σας συγχαίρω για τον διορισμό σας και θα ήθελα να αναφερθώ στα λόγια της κυρίας Ούρσουλα Φαντερ Λάιεν σχετικά με το 50% όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ποιο είναι το πρώτο συγκεκριμένο μέτρο που μπορείτε να μας αναφέρετε ως μέρος αυτής της δέσμης μέτρων. Και δεύτερον, στη δήλωσή της σχετικά με τη συμπερίληψη και της ναυσιπλοείας και της αεροπορίας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Πώς σκοπεύετε να το κάνετε αυτό, διότι είναι θέματα διεθνών μεταφορών όλες οι πτήσεις ε, που με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πληρώσουν τέλος ε, για το διοξίδιο του άνθρακα. Πώς σκοπεύετε να το κάνετε αυτό. Τρίτον, το θέμα της αποθήκευσης της ενέργειας. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι στον τομέα αυτών σχετικά με τα συστήματα αυτά, διότι από διάφορες υπηρεσίες της, προ... Επιτροπής. Ακούσαμε ότι η πράσινη ενέργεια χρειάζεται και κάποιες διασφαλίσεις ε, και η αποθήκευση θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο θέμα. Πώς το βλέπετε και ποιο πιστεύω ότι θα είναι το... ποια θα είναι η τιμή κατόφλη της κιλοβατόρας για να είναι βιώσιμο ένα τέτοιο σύστημα. Και μια ακόμα ερώτηση. Αναφερθήκατε στη στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Ήτρε. Αυτό το εκτιμούμε πολύ. Μας αρέσουν οι εκπλήξεις, ε, δεν μας αρέσει όμως να μας ευνηδιάζετε. Πιστεύετε ότι στο μέλλον θα μπορούμε να συμμετέχουμε στη διαδικασία κατάρτισης των νομοθετικών πράξεων, ώστε να γνωρίζουμε λίγο πιο νωρίς ε, ε, ποιοι είναι οι στόχοι σας. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον κανονισμό για το σύστημα εμπορίας εκπομπών και για την βιομηχανία χάλιβα είχαμε πολύ υψηλές τιμές. Πώς είναι δυνατόν να θέτουμε ένα σημείο αναφοράς πιο ψηλά από ότι το καλύτερο εργοστάσιο της Ευρώπης. Επευθύνθηκε λοιπόν σε εμάς η βιομηχανία χάλιβα και δεν θα θέλαμε τέτοιους ευνηδιασμούς στο μέλλον. Ελπίζουμε να μας θεωρήσετε εταίρους και σας ε, καλωσορίζω, στην, ε, σας συγχαίρω για την ε, ανάληψη της νέας σας θέσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Πέτερσεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτρέψτε μου και εμένα να σας συγχαρώ για την ανάληψη της νέας αυτής και πολύ σημαντικής θέσης. Φυσικά με ενδιαφέρουν πάρα πολύ την Επιτροπή μας, ε, τα σχέδια σας και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της εφαρμογής που ανέφερε και η, κυρία, και κυρία Καβάλιο, διότι δεδομένων των όσων υιοθετήσαμε στην προηγούμενη θητεία, δεδομένου του τεράστιου αγκουδουλιάς που έχει γίνει, η συζήτηση θα επικεντρωθεί γύρω από την εφαρμογή και πώς τα κράτη-μέλη θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. πώς μπορείτε λοιπόν να αναπτύξετε περαιτέρω τους προβληματισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα αυτό. Ξέρω ότι ναι, είναι πολύ διπλωματικό να λέτε ότι θα βοηθήσετε τα κράτη-μέλη. Μερικές φορές όμως χρειάζεται ίσως να λάβετε και πιο αυστηρά μέτρα για να διασφαλίσετε την σωστή εφαρμογή όλης της νομοθεσίας. Θα παρακαλούσα λοιπόν να αναπτύξετε λίγο το θέμα αυτό. Και τέλος, μια συγκεκριμένη ερώτηση. Αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, κάτι που σίγουρα όλοι θέλουμε, οι βιώσιμες πηγές ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να έχουν ακόμα υψηλότερη θέση στο χαρτοφυλάκιο αυτό και νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να ξανανοίξουμε την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεδομένης της ε, περαιτέρω πτώσης των τιμών στην ηλιακή και ολική ενέργεια. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, ε, το σκέφτεται και αυτό η Κομισιόν. Σας συγχαίρω και πάλι και προσβλέπω στην καλή συνεργασία. Ευχαριστώ κύριος Νινίστο. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την ανάληψη της νέας σας θέσης. Θα συνεχίσω στα αγγλικά, μην ανησυχείτε. Δεν μιλώ τόσο καλά δανέζικα. Φινλανδός είμαι. Σας συγχαίρω για την καινούρια σας θέση και προσβλέπω στην επόμενη πενταετία όπου τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα με τις παρούσες δεσμεύσεις δεν αρκούν για να πετύχουμε τους στόχους μας όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποδοτικότητα της ενέργειας. Υπάρχει λοιπόν σημαντικό κενό στα εθνικά σχέδια μέχρι στιγμής. Ε, πώς προβλέπετε εσείς να συνεργαστείτε με τα κράτη-μέλη και με τις κυβερνήσεις για να συμπληρώσετε το κενό αυτό. Και δεύτερον, ε, η υποψήφια πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σκοπεύει να ε, επανεξετάσει τους ε, στόχους και σε κάποιες χώρες οι στόχοι του 2050 θα μεταφερθούν στο 2035, για παράδειγμα και στη δική μου χώρα, τη Φιλανδία. Θα Έχουμε λοιπόν μια κλιματική πολιτική, όχι για τα επόμενα λίγα χρόνια, αλλά θα έχουμε έναν βιώσιμο δρόμο μέχρι το, 2015, μέχρι το 2050, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα του μεθανίου, τις εκπομπές. διότι το μεθάνιο είναι σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου, θα πρέπει να ασχοληθούμε με την αεροπορία, με ε, την ναυτιλία και με την ε, επιδότηση των ορυκτών καυσίμων. Η ομάδα μου φοβάται ότι... Θα εξετάσουμε ένα περιορισμένο φάσμα εργαλείων ε, για να πετύχουμε τους στόχους μας, παρακάμπτοντας σε κάποια άλλα πολύ σημαντικά, όπως είναι οι επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων. Πώς ε, το βλέπετε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σπόρκια. Σας ευχαριστώ. Και συγχαρητήρια για το διορισμό σας. Εγώ έχω να κάνω ε, μια ερώτηση σε σχέση με τις ε, περιφέρειες που ε, χρησιμοποιούν ακόμα άνθρακα. Θα ενθαρρύνεται για την βιομηχανική μετατροπή ή σκοπεύετε να ε, θέσετε σε εφαρμογή κοινωνικά μέτρα. Κύριε Κραζεντόφσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Έχω δύο ερωτήσεις αφορούν και ιδέες που ανέφερε η Ursula von der Leyen στην ομιλία της. Ανέφερε ένα ταμείο μετάβασης. Τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτό το ταμείο και έπειτα για το φόρο επί του άνθρακα. Ισχύει αυτή η ιδέα, θα δουλέψετε πάνω σε αυτή την ιδέα, σε αυτή τη θητεία. Και έπειτα αν μπορείτε να μας πείτε κάτι για το ποια είναι τα προγράμματα, τα σχέδια σε σχέση με το φυσικό αέριο. Γιατί ακούγονται φήμες ότι, το νέο, ότι θα προταθεί νέο νομοθετικό πακέτο από την Κομισιόν σύντομα. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε ή κάποιες κεντρικές ιδέες αυτού του πακέτου. και για την αναθεώρηση της οδηγίας ε, περί φυσικού αερίου. Ποια είναι η κατάσταση πρόοδου. Ε, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε. Σας ευχαριστώ. Okay. Euh, merci, Madame la Présidente. Félicitations. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, ο κύριος Μπομπά. Ε, ε, ευχαριστώ και συγχαρητήρια στη Γενική Διευθύντρια. Συγχαρητήρια, αλλά η δουλειά που έχετε να κάνετε είναι, το έργο σα είναι τεράστιο και πήγον, κατεπήγον. Το διαβάσατε και εσείς στην τελευταία έκθεση του ΖΙΕΚ που μας λέει πως αν θέλουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό θα πρέπει να καταφέρουμε να φτάσουμε το 2020 στο ανώτερο όριο εκπομπών αερίων ε, παγκοσμίω. Δυστυχώς ξέρετε ότι εδώ και τέσσερα χρόνια έχουμε ξαναρχίσει προς τα πάνω να πηγαίνουμε και το είπατε και εσείς ότι το 75% οφείλεται στην πολιτική ε, ενεργειακής παραγωγής, παραγωγής μάλλον ενέργειας. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε και να τηρήσουμε τους στόχους που έχουμε εμείς ήδη θεσπίσει αλλά ε, δυστυχώς είναι αυτό το μέχρι σήμερα παρκές. Ε, ε, ε θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το 2050 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιστημονικές εργασίες έχουν αποδείξει πως είναι δυνατό, είναι εφικτό. Εσείς θα δουλέψετε γύρω από αυτές τις επιστημονικές μελέτες ώστε να μπορέσουμε αύριο να αυξήσουμε και να υψώσουμε και πάλι τους στόχους μας. Ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you very much. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επειδή έχουμε αργήσει, θα σας δώσουμε την δυνατότητα να απαντήσετε τώρα σε ερωτήσεις των συντονιστών και μετά θα ακούσουμε όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους συντονιστές για τα καλά σας λόγια ε, και για τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ομαδικά γύρω από τα, τα διάφορα θέματα και να μην απαντήσω ε, μεμονωμένα στον καθένα από εσά άμεσα. Αλλά βέβαια, αν ε, απαντήσετε καταλήλως ή πλήρως, ε, μάλλον αν δεν απαντήσω πλήρως, θα σε επανέλθω. Να αρχίσουμε με τις ερωτήσεις που αφορούν την εφαρμογή. Είμαι ευτυχής που αρκετοί από εσά τονίσατε την εφαρμογή. Όπως είπα στις εγωγικές μου παρατηρήσεις, η εφαρμογή του νόμου είναι σημαντική για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θεσπίσει και πρέπει να εστιάσουμε στην εφαρμογή και να επιμείνουμε στην εφαρμογή γιατί δεν είναι κάτι το βραχυπρόθεσμο ε, για που αφορά μόνο τη μεταφορά του νόμου της οδηγίας, με συγχωρείτε, σε εθνική νομοθεσία, αλλά είναι κάτι το οποίο μονίμως θα πρέπει να παρακολουθείτε από τα κράτη-μέλη. Σκοπεύουμε να συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επίσης σε σχέση με την εφαρμογή ε, της νομοθεσίας και να σας ενημερώνουμε για την πρόοδο που ε, σημειώνεται. Τώρα, ε, τέθη το ερώτημα ε, συγκεκριμένα για τα εθνικά προγράμματα ενέργειας και κλίματος ε, και τα κενά που έχουν παρατηρηθεί σε κάποια κομμάτια στις εκθέσεις. Καταρχάς είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι είχαμε τα, σχέδια, τα εθνικά σχέδια πριν το καλοκαίρι και τη δυνατότητα να εξετάσουμε αυτά τα σχέδια και να επιστρέψουμε προς τα κράτη-μέλη με επικοδομητικά σχόλια. Και αυτό είναι ένα σημαντικό και χρήσιμο ε, βήμα ε, στη δικασία γιατί έτσι έχουμε χώρο ελιγμού πριν το τέλος και ε, στα τέλη του χρόνου από τότε που υποβάλαμε τα σχόλιά μας στα κρατημέλη είχαμε θετικά σχόλια. Νωρίτερα σήμερα η συνάδελφος Πάλι Βίνιο που είναι επικεφαλής της ε, μονάδας πολιτικής της DG Ενέργειας δουλεύει για αυτές τις προτεραιότητες και είδαμε πως υπάρχει η δέσμευση για την ε, ε, εξέταση αυτών των προτάσεων και των σχολείων που κάναμε. 24 Σεπτεμβρίου θα έρθω σε επαφή με τους Γενικούς Διευθυντές της Ενέργειας των Κρατών Μελών και βεβαίως έχουμε και διάφορες τεχνικές συνεδριάσεις που θα γίνονται συνεχώς και τακτικά ώστε να εξασφαλίσουμε πως ε, θα μείνει ζωντανή αυτή η δέσμευση και θα παρακολουθούμε και τις βελτιώσεις ε, ε, που γίνονται. Έγινε ερώτηση για τα ορυκτά καύσιμα και τις επιδοτήσεις και κατά πόσο αυτά έχουν αντιμετωπιστεί στα εθνικά σχέδια. Θα πρέπει, σύμφωνα με τους κανόνες, να υπάρχει ε, εντοπισμός των δεσμεύσεων για το ορυκτά καύσιμα που, ε, επιδοτήσεις που χορηγούνται και άρα αυτά, ε, αν δεν έχουν αναφερθεί στα σχέδια, στα προσχέδια μάλλον, απαιτούμε από τα κατημέλη να επανέλθουν και να μας πούν πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το θέμα. Ε, εν γέννη, οι τομεί τη επάρκεια, τη ενέργεια και των ανανεώσιμων πηγών απαιτούν περισσότερη φιλοδοξία αλλά και περισσότερε λεπτομέρειε ε, για τα μέτρα και τις φωτοβουλίες που σκοπεύουν να αναλάβουν τα κάτι μέλη. Και εδώ δουλεύουμε με τα κάτι συνεργαζόμαστε για να δούμε πώ θα προχωρήσουν. Υπάρχει και ένα πιο γενικό θέμα το οποίο ε, ετέθη για το πώς η εφαρμογή και οι νέες φιλοδοξίες θα, συνεργα... θα συνδυαστούν με τη νέα πράσινη συμφωνία, τη Green Deal. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε κανέναν από τους στόχους. Καταρχάς είχαμε τους στόχους του 2020 και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα τους στηρίσουμε αυτούς. Να εξασφαλίσουμε πως τα κράτη-μέλη και τα σχέδιά τους, τα εθνικά τους σχέδια ανταποκρίνονται σε αυτούς τους στόχους. Έπειτα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας στους στόχους του 2030 και όπως αναφέρατε στα ερωτήσει σας και τα σχόλιά σας ε, και συγκεκριμένα ο κύριος Νίκα το ανέφερε, η Ursula Leyen τόνισε την αύξηση στο 50% για το 2030 και ακόμα και περισσότερο ίσως. Άρα λοιπόν πρέπει αυτή η δουλειά να γίνει παράλληλα με την εκτίμηση των αξιολόγηση των σχεδίων, αλλά τα εθνικά αυτά σχέδια για την ενέργεια παραμένουν το βασικό εργαλείο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους του 20 και του 30 πρώτα. Συνετέθη μια ερώτηση και αυτό αφορά επίσης ε, την εφαρμογή για την οικονομία και την ανάγκη επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία. Πιστεύω πως ε, ο συσχετισμός με την οικονομία, την ανάγκη για μια δίκαιη μετάβαση, εξέταση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας, είναι και θα παραμείνουν κεντρική σημασία για τη διατύπωση των πολιτικών μας στο μέλλον. Αυτές οι πτυχές σαφώς και αναφέρονται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές από την ε, πρόεδρο, την υποψήφια της Επιτροπής και βεβαίω θα είναι αυτά τα πρώτα ίσω τα, πιο συγκεκριμένα μέτρα. Με βάση τι πολιτικέ κατευθυντήριες γραμμέ έχουμε μια καλή αλληλουχία που ε, να ξεκινήσουμε με την συμφωνία Green Deal μέσα στι πρώτε 100 μέρες και συνέχεια με κλιματική νομοθεσία καθώς και με το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση καθώς και την βιομηχανική πολιτική. Υπάρχει λοιπόν αλληλουχία για τις πρώτες 100 μέρες, αλλά και για το 2021, για τα προγράμματα, τους στόχους και ένα σωρό άλλα μέτρα που ε, αναφέρονται εκεί. Όπως είπα, δεν μπορώ να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα γίνουν όλα αυτά στην πράξη, γιατί είναι πολιτική απόφαση που θα πρέπει να λάβουν οι ε, νέοι επίτροποι. Στο πλαίσιο αυτό, μια από τις ερωτήσεις αφορούσε το σχέδιο εμπορίας εκπομπών τι κάνουμε λοιπόν με τις ε, αεροπορικές μεταφορές και τις υποδείξεις ε, της υποψήφιας ε, προέδρου στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές αλλά και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Ευρωκοινοβουλίου και πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε τους στόχους. Τέθη συγκεκριμένη ερώτηση σε σχέση με τον τομέα του Χάλιβα και το, ενός, μιας χαλιβουργίας που δεν απέχει και πολύ από εδώ. Στι πολιτικέ κατευθυντήριε γραμμές, η υποψήφια πρόεδρος για τις αεροπορικές μεταφορές αναφέρθηκε στην ε, δωρεάν ε, εκχώρηση ε, ποσοστώσεων και στη μείωση αυτών σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα. Και αυτό είναι κομμάτι των θεμάτων που θα πρέπει να εξετάσει η νέα Επιτροπή μόλις αναλάβει καθήκοντα. Ετέθη ερώτηση για τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας, για το κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας και αν πρέπει να κάνουμε και περισσότερα ή αν πρέπει να αναθεωρήσουμε την νομοθεσία. Να υπάρχει ρήτρα αναθεώρησης της νομοθεσία μας. Θα δούμε φυσικά σε ποιο βαθμό και πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Θα συνεργαστούμε στενά και θα ε, ε, διαβουλευτούμε με το Ευρωκοινοβούλιο στο πλαίσιο αυτό με βάση τα όσα θεσπίστηκαν. Πιο γενικά και επανέρχομαι στο θέμα της συμμετοχής του Ευρωκοινοβουλίου στην νομοθετική διαδικασία, πιστεύω πω η υποψήφια πρόεδρο στι πολιτικέ τη κατευθύνσει ε, δήλωσε σαφώ προθέσει να ενισχύσει τη συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο, να δώσει ισχυρή ρόλο στη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υποβολή, στην πρόταση για ε, ε, νομοθεσίε και αναφέρθηκε στη δυνατότητα του, να δράσει το Κοινοβούλιο στην υιοθέτηση ψηφισμάτων που προτείνει, θα προτείνουν στη Κομισιόν να ε, εκπονήσει νομοθεσία. Αυτά όλα νομίζω αναφέρονται σαφώς στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές. Και στα επόμενα χρόνια θα συνεργαστούμε για την εφαρμογή όλων αυτών μετά από τη σαφή δέσμευση της υποψήφιας Προέδρου για ισχυρότερη συνεργασία, στενότερη συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο. Σε σχέση τώρα με την έρευνα και την καινοτομία, υπήρξε το ερώτημα για την αποθήκευση ως ένας από τους τομείς που πρέπει να βελτιώσουμε την τεχνολογία μας. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που αφορούν στην αποθήκευση. Και ένα συγκεκριμένο σημείο που εξετάζουμε είναι αυτό της ενσωμάτωσης του τομέα. Με άλλα λόγια, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές πηγές ενέργειας που να αλληλοσυμπληρώνονται αλλά και να μετατρέψουμε, να έχουμε ηλεκτρική ενέργεια σε υδρογόνο ή και σε άλλες πηγές ενέργειας. Είναι ένα σύνδεσμο μεταξύ διαφορετικών τομέων και αυτό είναι κάτι που θα είναι σημαντικό για μας τα, επόμενα χρόνια, είναι κάτι πάνω στο οποίο εργαζόμαστε και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όταν σχεδιάζουμε α, την έρευνα και την καινοτομία. Νομίζω ότι αν κάτι είναι σαφές είναι ότι υπάρχει ανάγκη για χρηματοδότηση, υπάρχει ανάγκη για επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία και αυτό θα πρέπει βεβαίως να είναι ε, μέρος του PDP αν θέλουμε να παραμείνουμε σε μια ηγετική θέση σε ό,τι αφορά την καθαρή ενέργεια και την καθαρή βιομηχανία. Αν η Ευρώπη θέλει να επανέλθει σε ηγετική θέση σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν αναφέρομαι στις επενδύσεις και την επιχορήγηση, αναφέρομαι τόσο σε δημόσιο όσο σε ιδιωτική. Μίλησα για το πολιετές δημοσιονομικό πρόγραμμα, αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις. Ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όταν έχουμε χρηματοδοτήσει, τότε είναι βιώσιμα τα προγράμματα αυτά και θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας. Υπήρξε και ένα ερώτημα σχετικά με πιθανές πρωτοβουλίες που αφορούν το φυσικό αέριο και την οδηγία για το φυσικό αέριο και πώς αυτή έχει γίνει αποδεκτή από κάποιες αγορές. Πιο συγκεκριμένα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη οδηγία με τις πρόσφατες τροπολογίες της που διασαφηνίζουν τον τομέα, το πεδίο δράσης της οδηγίας είναι σαφές πλέον ότι αναφερόμαστε στην ευρωπαϊκή περιοχή. Είναι συμβατή η οδηγία αυτή τόσο με τις Συνθήκη της Ένωσης όσο και με τις ε, διεθνείς δεσμεύσεις μας. Επομένως, σε ό,τι αφορά την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα βρεθούμε εκεί με αυτοπεποίθηση και βεβαίως θα υπερασπιστούμε της οδηγίας για το φυσικό αέριο. Όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά και ε, σε οποιαδήποτε διαμάχη μπορεί να προκύψει. Δεν είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε με το χρόνο μας, αλλά βεβαίως και είμαστε διατεθειμένοι να απαντήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το φυσικό αέριο και μια πιθανή μελλοντική πρωτοβουλία, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να ενσωματώνουμε το φυσικό αέριο στη μετάβασή μας, στην ενεργειακή μας μετάβαση. Είναι μια πηγή ενέργειας που είναι πολύ σημαντική για την ενεργειακή μας μετάβαση. Είναι ανάγκη να εξετάσουμε με ποιο τρόπο θα το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τις εκπομπές άνθρακα, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία που έχουμε ε, με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό είναι κάτι που θα χρειαστεί καινοτομία, θα χρειαστεί τεχνολογία, θα χρειαστεί επενδύσεις. Έχουμε όμως αρκετά εργαλεία για να το κάνουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά μια ενδεχόμενη πρωτοβουλία για το φυσικό αέριο, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τοποθετήσουμε τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες τόσο στα πλαίσια της μετάβασης που διανύουμε αυτή τη στιγμή, όσο και στα πλαίσια του Green Deal, ούτω ώστε να έχουμε και φτηνή ενέργεια. Το ερώτημα αυτό και πάλι είναι ένα πολιτικό ερώτημα και δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Μπορώ να σας πω όμως ότι είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε τόσο στα πλαίσια της απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα και της μετάβασης. Πιστεύω ότι έχω απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που εγείρατε και αν μου ξέφυγε κάτι θα χαρώ να επανέλθω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, τώρα έχετε το λόγο. Ένα λεπτό καθένα σας. Τα μέλη της Επιτροπής. Η κυρία Ντεκαστήλιο έχει το λόγο πρώτη. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω ισπανικά. Συγχαρητήρια για τον διορισμό σας. Και είναι χαρά μας που βρίσκεστε εδώ. Έχετε μεγάλη εμπειρία σε πολλούς ε, τομείς της Κομισιόν και από όσο γνωρίζουμε είσαστε ακούραστοι και ε, πολύ νυφάλιος άνθρωπος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, περάσαμε από την προηγούμενη θητεία της απόφασης στην θητεία της εφαρμογής. Η νομοθετική προσπάθεια έγινε στην προηγούμενη θητεία και τώρα έρχεται η προσπάθεια της εφαρμογής όλων αυτών. Και δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος, πρέπει να ε, τα εφαρμόσουμε. Ε, μπορεί να κάνει κανείς λάθος από υπερβολή ή από λάθος, γιατί μπορεί να θέλει πολλά δηλαδή και να μην είναι ή μπορεί να κάνει λάθος στην εφαρμογή. Εμείς έχουμε λοιπόν πολύ λεπτομερή νομοθεσία όσον αφορά το σεθνικό προπολογισμού των κρατών μελών. Εκεί πάντοτε δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες. Πάντοτε ξέρει κανείς ε, αν θα επιτύχει ή αν θα αποτύχει στην επίτευξη του ελλείμματος και πότε και γιατί. Θα πρέπει τέτοιο σύστημα να εφαρμόσουμε και για τα εθνικά σχέδια για ε, την ενέργεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή την εμπειρία που έχουμε από τα εθνικά ε, σχέδια για το προπολογισμό για να κάνουμε ρεαλιστικά ε, πλάνα και να μην αποτύχουμε και έπειτα. για τις εκπομπές της βιομηχανίας είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πώς θα γίνει η διακοπή της χρήσης του άνθρακα. Ε, γιατί αυτή έχει τεράστιο αντίκτυπο στις εκπομπές της βιομηχανίας και κατά συνέπεια για την οικονομία. Αλλά κυρίως το πρώτο κομμάτι, δηλαδή, αυτό που ανέφερα, Δε από την απόφαση, την νομοθετική στην εφαρμογή πρέπει να περάσουμε και είναι πολύ σημαντικό να τα καταφέρουμε και μπορείτε να βασίζεστε στην υποστήριξη μας. Ευχαριστώ συνάδελφοι, ξέρω πως είναι δύσκολο να μην έχετε χρόνο. Είναι όμως τόσο πολλά που θέλουμε να πούμε με την Γενική Διευθύντρια και πιστεύω ότι θα έχουμε ευκαιρίες στο μέλλον. Επομένως, σας παρακαλώ πολύ να σέβεστε το χρόνο. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριε Ζωρίνιο, θέλω να σας ε, συγχαρώ για τον διορισμό σας. Εγώ ήμουν σκιώδης συζητητή στους σοσιαλιστές για την κανονισμό, για την διακυβέρνηση, για την ενεργία και έχω συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα σχέδια ενέργεια ε, κλίματος ως πολιτική δέσμευση και ως μέσο για τους πολίτες. Πολιτική ε, ε, δέσμευση. Έχουμε το καλό νέο του πράσινη συμφωνία του Green Deal, αλλά έχουμε το ανησυχητικό ζήτημα ότι τα σχέδια τα εθνικά δεν φτάνουν τους ε, σημερινούς ισχύοντες στόχους. Πώς θα αποφύγουμε λοιπόν το να, αντί να επιταχυνθεί η διαδικασία να έχουμε δύο πλαίσια που τελικά μπορεί να το φρενάρουν. Έπειτα, για τους πολίτες, όπως σας είπα, είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να συμμετέχει στην συζήτηση για την ενέργεια. Στην Πορτογαλία έγινε εξαιρετική συζήτηση, αλλά με τους ειδικού. Πρέπει να πάμε κοντά στους πολίτες, να μην μείνουμε μόνο στη συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες. Προβλέπεται στον κανονισμό η ε, δημιουργία ε, πλατφορμών των πολιτών για την επικοινωνία με τους πολίτες. Πώς σκοπεύετε να στήσετε αυτές τις πλατφόρμες. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μιχαήλοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια, κύριε Γενική Διευθυντρία. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και κάθε επιτυχία σε αυτό το δύσκολο τομέα πάνω στον οποίο θα εργαστείτε. Κρατώντας κατά νου τον πολύ ευγενικό τρόπο που μας ενημερώσατε, για τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, θα σας ζητήσω να είστε πιο συγκεκριμένοι. Πιστεύετε ότι έχετε αρκετά όργανα, αρκετά εργαλεία για να μπορέσετε να επηρεάσετε τα κράτη-μέλη όταν προετοιμάζουν τα εθνικά του σχέδια. Δυστυχώς, ε, όταν είχαμε τα, τα προσχέδια δεν είχαμε και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά σχόλια. Για παράδειγμα, έλλειψη φιλοδοξίας και ιδιαίτερα σαφή μέτρα. Πιστεύετε ότι έχετε αρκετά όργανα για να μπορέσετε να ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη, να κατευθύνετε τα κράτη-μέλη για να ε, έχουν ε, μέτρα μεταξύ των ε, διαφόρων τομέων, όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπούζεκ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να συμφωνήσω και εγώ με τους συναδέλφους, να σας συγχαρώ για την καινούρια θέση σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, διαθεσιμότητά σας εμάς εδώ να δώσετε το παρόν. Όπως ορθά είπατε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή παλαιότερων νόμων που υιοθετήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Από την οπτική γωνία όμως της ε, Ενεργειακής Ένωσης έχουμε τους πέντε πυλώνες μας. Για να κρατήσουμε λοιπόν την ισορροπία μεταξύ των πυλώνων αυτών που είναι πολύ σημαντική. Για παράδειγμα για την έρευνα και την καινοτομία και εσείς ίδια κάνατε λόγο. Όμως την εξασφάλιση της προμήθειας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι αντικρουόμενα τα δύο αυτά στοιχεία, αλλά σε κάποια κράτη-μέλη μπορεί και να είναι αντικρουόμενα. Πώς, ε, τι μπορείτε να προτείνετε για το, για το πρόβλημα αυτό. Χρειαζόμαστε στήριξη για την ενσωμάτωση γενικότερα, εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Θα ήθελα να, να δω κάποια τέτοια πρόταση για τις ε, περιφέρειες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε το σήμα, να περάσουμε το μήνυμα στους πολίτες μας ότι είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπρούκνερ τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλήσατε για αποθήκευση της ενέργειας και υποστηρίχθηκε ότι δεν υπάρχει ακόμη κάποια κατάλληλη λύση για την αποθήκευση της ενέργειας. Ε, όμως υπάρχουν μεγάλες τεχνικές εγκαταστάσεις που όμως ε, δεν λειτουργούν εμπορικά, διότι εν μέρη, στη Γερμανία τουλάχιστον, ε, πρέπει να πληρώνουν διπλά τέλη. Ε, τέλος για το ηλεκτρικό ρεύμα και τέλος για την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Και γι' αυτό δεν συμφέρουν σε σχέση με τον άνθρακα. Ε, αλλά αυτό είναι πολιτική βούληση. Δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε τη χρήση ε, του λιθάνθρακα τόσο γρήγορα. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει για να εξαλείψουμε τέτοια παράλογη εθνική νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χάσελ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και από μένα στη Γενική Διευθύντρια για την ε, ανάληψη των καθηκόντων της. Ε, σας εύχομαι και εγώ κάθε επιτυχία. Έχω δύο σύντομα ερωτήματα. Αναφερθήκατε κυρίως ως προβληματικό σημείο ε, στα σχέδια αυτά, στην επάρκεια της ενέργειας, ό,τι αφορά τα εθνικά σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια. Τι πιστεύετε ε, για την άποψη που εκφράστηκε από μερικούς που επιμένουν σε μια αύξηση ανανεώσιμης ενέργειας και πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει σε κάποια κράτη-μέλη μόνο αν χρησιμοποιούσαμε ένα σύστημα επιδοτήσεων αυξάνοντας την τιμή για τη χρήση του φυσικού αερίου, ιδίως για τα νοικοκυριά, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση της, των συνθήκων φτώχειας, ιδίως στην Κεντρική Ευρώπη. Και το δεύτερο ερώτημά μου, τι βλέπετε ως προοπτική σε ό,τι αφορά τα ορυκτά καύσιμα και πιο συγκεκριμένα τον άνθρακα. Αν αντικατασταθεί, αν πιστεύετε θα αντικατασταθεί από την κατανάλωση φυσικού αερίου, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σπυράκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύρια Πρόεδρε. Συγχαρητήρια και στη Γενική Διευθύντρια. Επιτρέψτε μου να επιμείνω στα βασικά, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε αν σύμφωνα με την ε, Ursula von der Leyen. Χρειαζόμαστε επιπλέον νομοθεσία, ούτως ώστε να έχουμε μια καινούρια, ένα καινούριο Green Deal ή αν απλά πρέπει να εφαρμόσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία και να προσθέσουμε εδώ και εκεί κάποια νέα κομμάτια νομοθεσίας, δευτερευόντως κάτι που αφορά συγκεκριμένα την Ελλάδα. Γιατί όπως ξέρετε αντιμετωπίζουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και έχουμε πολλές ε, δυνατότητες, περίπου 600 εκατομμύρια. Θα ξεκινήσετε με την ελληνική κυβέρνηση ένα καινούριο σχέδιο που να αφορά στο PPC. Ξέρετε ότι άπτεται τη εθνική μα αρμοδιότητα, αλλά οπωσδήποτε θα χρειαστούμε και τη βοήθεια τη Επιτροπή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τομπισόφσκι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πολύ να ακούσω λίγα λόγια από σας σχετικά με τις ε, περιοχές εξόρυξης άνθρακα της Ευρώπης. Πρέπει να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης στις περιφέρειες αυτές που θα αντικαταστήσουν τις ε, θέσεις εργασίας που χάνονται. Επίσης, έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να καλύψουμε το κόστος αυτό και να έχουμε όφελος από την ενεργειακή μετάβαση στην Πολωνία, στην Τσεχία και την Ρουμανία. Επίσης, ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε μία ερώτηση που τέθηκε. Αναφερθήκατε στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. και την πρόταση για αύξηση του τέλους ε, για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ένα τέτοιο τέλος μπορεί να οδηγήσει σε προστασία των δικών μας παραγωγών ε, στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Έχετε προβληματιστεί πάνω στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Γκάιερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ. Η δική μου ερώτηση έχει σχέση με τη σχέση ανάμεσα στους διάφορους τομείς η συνεργασία μεταξύ διαφόρων βιομηχανικών τομέων μπορεί να μας ε, βοηθήσει ε, στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Ε, δεν άκουσα τίποτα σχετικό με αυτό και επίσης δεν έχω αρκετή φαντασία να σκεφτώ πώς θα το πραγματοποιήσετε αυτό. Υπάρχει, υπάρχουν ευκαιρίες όμως, υπάρχουν δυνατότητες με, την, με, τον, με τη συνεργασία ανάμεσα σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Θα ήθελα παρακαλώ να ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Ε, ο κύριος ε, Φλέγκος, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Προσλέπω στην καλή συνεργασία μας στο μέλλον. Εγώ ήθελα να αναφερθώ στην εφαρμογή της νομοθεσίας, κάτι που ανέφεραν διάφοροι συνάδελφοι. Ναι, γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν συνεργαστεί στην κατάρτιση των ενεργειακών του σχέδιων. Ε, κάποια κράτη-μέλη ήταν πιο φιλόδοξα, αλλά λιγότερο. Η δική μου ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Η Ευρωπαϊκή Επίτροπη θα μπορούσε να αξιολογήσει συγκεκριμένα και αντικειμενικά τα προγράμματα αυτά, να διαπιστώσει αν υπάρχουν προβλήματα και να κινητοποιήσει όλα τα κράτη-μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξή τους. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, εξετάσει το ενδεχόμενο ποινή στα μη αρκετά φιλόδοξα σχέδια. Ε, και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ. Όσοι συζητήσει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, δεν με εκπλήσει το χάσμα όσον αφορά τις φιλοδοξίες των κρατών μελών, διότι ε, ήταν ε, πολύ διστακτική όσον αφορά την ε, αρχική αύξηση των στόχων. Επίσης, δίσταζαν να επιτρέψουν στους καταναλωτές να παράγουν τη δική τους ενέργεια. Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων νομίζω θα είναι υψής της για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμμετείχα σε διάφορες εκδηλώσεις πάνω στα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και διάφοροι άνθρωποι μου είπαν ότι αν υπήρχε η ότι ήθελαν να παράγουν τη δική τους ενέργεια, αλλά υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο. Μήπως θα μπορούσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας ε, διετούς εκθέσεως ε, που να διαπιστώνει την πρόοδο στον τομέα αυτών και τα λάθη που θα πρέπει να διορθωθούν. Διότι θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα των ε, ποινών και των αμοιβών. Ευχαριστώ κύριε Τουσάν, παρακαλώ. Je vous remercie et j'adresse euh, également mes félicitations à Madame Jorgensen. Euh, les énergies fossiles... Θέλω και εγώ να συγχαρώ την κυρία του Γιόνσεν και τα ορυκτά καύσιμα είναι ακόμα ε, καταστροφικά όσον αφορά ε, την, το κλίμα. Τα, περιμένουμε ακόμα απόφαση από τα κράτη-μέλη. Πέρυσι μας είπαν 55 εκατομμύρια ε, ευρώ επενδύονται ετησίως σε αυτές τις επικίνδυνες, τα επικίνδυνα ενέργειας. Όμως κάποια κράτη-μέλη όπως και η Γαλλία ισχυρίζονται πως δεν χρηματοδοτούν πια τις τις ορυκτές πηγές ενέργειας, όταν αυτό είναι, είναι ψέμα. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε για να ε, αναγκάσετε αυτά τα κράτη να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους όσον αφορά τις άμεσες και έμεσες ε, επιδοτήσεις και πώς θα επιτύχετε το στόχο ε, της πάυσης κρίσης αυτών των ειδών ενέργειας μέχρι το 2050 για όλα τα κάτι μελη της Ένωσης. Thank you very much. Ο κύριος Φουλουκλάν. Ευχαριστώ πολύ. Να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, τα ενέζικα. Σας συγχαίρω για τον διορισμό σας. Ε, θα ήθελα να θέσω ερώτηση σχετικά με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις τιμές ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνεχώς υπερεκτιμούσε την τιμή πώληση της ανανεώσιμης ενέργειας. Και το, η τιμή αναφοράς για τις ηλιακές κυψέλες ε, είναι υψηλότερη από ό,τι για το 2030. Το ίδιο ισχύει για την αιωλική ενέργεια. Ε, έχουμε φτηνότερη ενέργεια αιωλική ε, από ότι οι τιμές αναφοράς ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις και θα ήθελα να ε, σε ρωτήσω αν σκοπεύετε να αλλάξετε πολιτική στον τομέα αυτών. Ε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπελαμή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ανάληψη της θέσης σας αυτή. Να μιλήσω κι εγώ γαλλικά και να σας κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, κυρίως ό,τι αφορά την υδροηλεκτρική ενέργεια. Όπως ξέρετε η Επιτροπή εδώ και αρκετά χρόνια ασχολείται με τον ανταγωνισμό για πάνω στον τομέα αυτό της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ένας τομέας που σήμερα παράγει μια ενέργεια παντελώς πράσινη αλλά πολύ πιο ακριβή. Ποια είναι η θέση σας πάνω στο ζήτημα αυτό. Δεν πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την συγκεκριμένη αυτή ενέργεια που μπορεί να μας εγγυηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια παντελώς καθαρή ενέργεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βάις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σε συγχαίροντείτε. Πολλές καλές ερωτήσεις ε, τέθηκαν σήμερα και θα ήθελα να συμφωνήσω με τον ε, συμπατριώτη μου Νίλς για το θέμα των δεδομένων σχετικά με τις τιμές της ενέργειας. Αλλά θα πρωτοτυπήσω, θα θέσω μια άλλη ερώτηση σχετικά με την επικοινωνία κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, την ενεργειακή μετάβαση που περνάμε, διότι έχουμε πολλές ψευδείς ειδήσει, ε, πολλά ψευδή δεδομένα, έχουμε ε, δημόσια στηλίτευση και δεν θα πρέπει μόνο η ΜΚΟ να αναφέρονται όταν μιλάμε για διάφορες ομάδες ε, συμφερόντων ε, στην Ευρώπη. Ε, θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, θα τα καταφέρουμε, θα πρέπει όμως να είμαστε και σαφείς όσον αφορά τις συστηματικές απειλές για τα συστήματα επικοινωνίας εντός της Ευρώπης. Πώς το βλέπετε λοιπόν αυτό και μήπως ε, θα, ε, θα πρέπει να υπάρχει διατομεακή προσέγγιση, να συνεργαστείτε για παράδειγμα με τη Γενική Διεύθυνση ε, Επικοινωνίας. Ευχαριστώ. Κύριος Γκονζάλης Κασάρας, παρακαλώ. Συγχαρητήρια κυρία Γιόγκερσεν για το διορισμό σας. Στην θέση αυτή έχετε δύσκολο ρόλο αλλά μεγάλη πρόκληση μπροστά σας και πολύ συναρπαστικό το θέμα σας θα πρέπει να δούμε πως το 2023 θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε τους ε, στόχους. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2023 μετά από τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις ε, που ανέλαβε η Ούρσονα Βαντελάγεν και έπειτα μιλάτε για τη δίκαιη μετάβαση. Εγώ προέρχομαι από τη Γαλλικία, μια περιοχή που και που κινητοποιείται γιατί καταλαβαίνει πως πρέπει να αλλάξει από τον άνθρακα. Έφτιαξε ε, μία ε, και το έχει κάνει, επενδύονται διαρκώς χρήματα, αλλά κάθε φορά έχουμε, έχει να αντιμετωπίσει ε, μεγαλύτερες απειλές. Τι μήνυμα μπορείτε να στείλετε λοιπόν από την Κομισιόν ώστε να εμπιστευτούν αυτή τη δυνατότητα δίκαιης μετάβασης. Υπάρχουν κέντρα απασχόλησης όπως αυτός ο σταθμός και αλλού στην Ευρώπη που θα επηρεαστούν. Επίσης, τι μέτρα έχετε σκεφτεί να, ε, να, να εφαρμόσετε όσον αφορά την ενεργειακή επάρκεια. Κυρία Παύλος. Merci. Ευχαριστώ και εγώ από πλευρά μου να συγχαρώ τη Γενική Διευθύντρια. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά σχέδια, καταλαβαίνω την προσέγγιση σας για τη συνεργασία. Παρ' όλα αυτά, 11 κράτη-μέλη ακόμη δεν έχουν δηλώσει μια κάποια ημερομηνία για στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για τους στόχους που έχουμε θέσει για την κλιματική αλλαγή. Τι πρόοδο έχετε κάνει στο τομέα αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, Επίσης, η φιλοδοξία για τους στόχους του 2050 αλλά και για τους στόχους που τέθηκαν στην Συμφωνία του Παρισιού θα αλλάξετε ίσως από ένα χρονικό πλαίσιο σε ένα σενάριο προϋπολογισμού. Το ερώτημα είναι πόσο άνθρακα εκπέμπουμε. Όχι μέχρι ποιο έτος θα, θα συνεχίσουμε να τον εκπέμπουμε. Το ερώτημα αυτό έχει εγερθεί αρκετές φορές. Όλες οι χώρες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Δεν πιστεύετε κι εσείς ότι είναι μια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μια ηγετική θέση στον τομέα αυτό της ε, καθαρής ενέργειας. Και άλλη μια ερώτηση. Συγγνώμη, έχετε εξαντλήσει το, χρόνο σας, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Κονκουλανάτρη. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Καλή τύχη στη δουλειά σας και καλή συνεργασία για τα επόμενα πέντε χρόνια. Πίστευω ότι δεν υπάρχει χρόνος για καινούριε ερωτήσεις. Να ρωτήσω λοιπόν και εγώ για τις μπαταρίες και για την αποθήκευση, γιατί υπάρχει νομοθεσία και θέλουμε βεβαίως να απαλλαγούμε από τις εκπομπές και ξέρουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία. Υπήρχαν φιλόδοξοι στόχοι και ιδέες από πλευράς της Επιτροπής. Είστε διατεθειμένοι να συνεχίσετε πάνω σε αυτό το δρόμο Ποιο είναι το μήνυμά μου. Συντονισμός, συντονισμός, συντονισμός. Να αναφερθούμε και στην ομιλία της Φόντερ Λάιν που έκανε λόγο για την ε, φορολογία. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται μεγάλη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Τόσα, τόσα σημεία θίξαμε, αλλά όχι αυτό. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά σχέδια τώρα, ο τομέας των κατασκευών Επίσης θα πρέπει να, θα πρέπει να συντονίσουμε ούτως ώστε να γίνει ευκολότερο για τα κράτη-μέλη να καταθέσουν τα, τα σχέδια αυτά. Ευχαριστώ. κυρία Καρβάιο. Ο κύριος Έλερ μάλλον μέσω της κυρίας Καρβάλιο. Δύο ερωτήματα θα σας ρωτήσω εκ μέρους του κυρίου Έλερε. Απλά ερωτήματα. Συνεργείς μεταξύ του προγράμματος Horizon Ευρώπη και του Ταμείου για την Καινοτομία. Μπορεί να υπάρξει μια συνεργία. Για παράδειγμα, την απαλλαγή από τις εκπομπές του άνθρακα. Δεύτερο ερώτημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για περιφέρειες οι οποίες εξαρτώνται από τον άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τόρια τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια σε Διευθύντρια και από δική μου πλευρά και για την σαφήνεια με την οποία μας παρουσίασε το σημερινό πλαίσιο ε, των προοπτικών. Θέλω να περάσω σε πολύ συγκεκριμένα αλλά σημαντικά ερωτήματα για τις διάφορες χώρες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων από πλευρά κάποιων κρατών μελών και το κατά πόσο το ε, επέτυχαν ή όχι και ρωτηθήκατε αν θα, ποια θα είναι τα μέτρα που θα επιβάλλετε. Κάποια κράτη θέλουν να κάνουν ένα πασάλιμα και να απλαπλώσουν τις καθυστερήσεις και εις βάρος των ε, χωρών οι οποίες τήρησαν τις ε, προθεσμίες. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει, θα, θα αντιτεθεί η ε, Κομισιόν. Δεν είναι κάτι το οποίο οδηγεί στην ανάληψη ευθυνών. Έπειτα, ολόκληρο το πρόγραμμα για τα ε, οικολογικά συμβατά ε, προγράμματα η Κομισιόν δεν το ενέκρινε, αλλά αυτό είναι μεγάλο ε, πλήγμα, γιατί οι παραγωγοί ηλεκτρικών συσκευών περιμένουν την έγκριση αυτή. Έπειτα, η συνδυασμός ανάμεσα στη εμπορικά στάνταρ και κλιματικά στάνταρ. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρία, ο κύριος Ευχαριστώ και συγχαρητήρια κυρία Γιόγκερσεν. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Εγώ προέρχομαι από τη νέα γενιά και βλέπω ε, την ε, ε, κατάσταση βρισκόμαστε στο χείλος καταστροφής, της καταστροφής. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που μπορεί να ληφθούν για να εφαρμοστεί το 55% για παράδειγμα στον τομέα της, ε, των κτηρίων και ε, ας πούμε μιλήσαμε και για την εξάλληψη της χρήσης του άνθρακα. Πώς θα βοηθήσετε ώστε τα κράτη-μέλη που δεν είναι ακόμα τόσο πεπισμένα ότι αυτό χρειάζεται και ότι επιφέρει πολλά ωφέλη όσον αφορά την υγεία, η οικονομία είναι, είναι πιο προσιτό, οθεί τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τα λοιπά. Πώς βλέπετε, μάλλον ποια είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα για σας αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Είμαι απολύτως βέβαιη ότι οι συνάδελφοι αν είχαν περισσότερο χρόνο θα είχαν θέσει ακόμα περισσότερες ερωτήσεις, αλλά εν πάση πτώση ας κάνουμε μια προσπάθεια να απαντηθούν κάποιες από τις ερωτήσεις τους τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους και πάλι για το θερμό καλωσόρισμα και τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις σας. Ε, χαίρομαι που δεν βλέπετε τις σημειώσεις μου, διότι ε, δυσκολεύομαι όλο και περισσότερο να διαβάσω τα ορνηθοσκαλίσματά μου. Θα κάνω όμως ό,τι μπορώ για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Θα τις ομοδοποιήσω στο βαθμό που είναι δυνατό και ελπίζω να επιδείξετε υπομονή ε, όσον αφορά τις ερωτήσεις που δεν θα απαντήσω ή που δεν θα απαντήσω αρκετά σαφώς ε, και θα προσπαθήσω να τις απαντήσω την, στην επόμενη φορά στην επόμενη συνάντησή μας. Αρκετοί από εσά ε, μίλησαν για τη συμμετοχή των πολιτών και την ε, σωστή επικοινωνία μαζί τους, να φροντίσουμε να μην υπάρχουν ψευδείς ειδήσει, fake news και να συμμετέχουν οι πολίτες στη δουλειά μας. Ε, ας ξεκινήσω από αυτό, διότι νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι το βασικό θέμα που μας ενδιαφέρει. τα τελευταία χρόνια. Είδαμε σημαντική συμμετοχή των πολιτών σε διάλογο, σε φόρουμ. Ε, στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, βλέπουμε σημαντική παρουσία των πολιτών ενδιαφέρον για τα κλιματικά θέματα και νομίζω ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε με βάση τα όσα ήδη έχουμε πετύχει και να συνεχίσουμε την ε, στενή επικοινωνία μας με τους πολίτες. Κάποιοι από εσά ε, τόνισαν ότι δεν είναι οι ίδιε οι θέσει σε όλη την Ευρώπη, σε όλε τι χώρε, σε όλου του τομεί, σε όλε τι γενιέ. Ε, φροντίζουμε όμω ε, να αφουγκραζόμαστε, να ακούμε όλου, να ακούμε τι ανησυχίε του και Διαβάζοντας τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Προέδρου Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ε, θα βρείτε αναφορά σε διάφορους παράγοντες της κοινωνίας μας, σε συμμετοχικές διαδικασίες, χώρες, περιφέρειες, βιομηχανικούς τομείς, ε, την κοινωνία των πολιτών, ε, νέους και ηλικιωμένους και νομίζω ότι αυτό είναι το ξεκίνημα μιας σημαντικής διαδικασίας επικοινωνίας και ελπίζω να μπορέσω να συμβάλλω και εγώ στη διαδικασία αυτή. Πιστεύω ότι και εσείς, ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως άμεσα εκλεγμένοι από τους πολίτες, θα παίξετε ε, ζωτικό ρόλο στα επόμενα χρόνια. Αρκετοί από εσά αναφέρθηκαν στους διαφορετικούς πυλώνες ε, της Ενεργειακής Ένωσης. Μας ενδιαφέρει το κλίμα, μας ενδιαφέρει η βιώσιμη και καθαρή ενέργεια. Υπάρχουν όμως και άλλοι τομείς τους οποίους θα πρέπει να προσέξουμε και ελπίζω να ήμουν αρκετά σαφής όταν σας ανέφερα την ε, δέσμευσή μας, ε, την αφοσίωσή μας ε, στους στόχους, μας ενδιαφέρει ο ρόλος του φυσικού αερίου στο πλαίσιο αυτό. Ως τμήμα της πράσινης μετάβασης, καθώς και η εγκατάλειψη της εξόριξης άνθρακα αναφέρθηκαν τα εθνικά σχέδια. Αναφέρθηκε ότι όχι όλα τα κράτη-μέλη ήταν σαφή ως προς τις προθέσεις τους. Αναφέρθηκε επίσης ότι τα ε, σχέδια για το κλίμα δεν είναι όλα απόλυτα σαφή όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα. και τέθηκαν και ερωτήσεις σχετικά με το τι θα κάνουμε τελικά στην πράξη εάν δεν αρκούν τα εθνικά σχέδια, εάν δεν ε, μας επιτρέπουν να πετύχουμε τους στόχους μας και αν δεν είναι αρκετά συγκεκριμένα. Να κάνω λοιπόν πρώτα κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Τα σχέδια που λάβαμε το καλοκαίρι ήταν σχέδια, ήταν προκαταρκτικά σχέδια, είναι ένα ενδιάμεσο ε, στάδιο που μας επιτρέπει να εξετάσουμε τα σχέδια αυτά και να επανέλθουμε με συγκεκριμένες παρατηρήσεις στα κρατη Όλα τα κρατη έχουν λάβει παρατηρήσεις και συστάσεις. Κάποια βρίσκονται πιο κοντά στους στόχους από ό,τι άλλα, αλλά ήδη έχουν επιτύχει τους στόχους του 2020 αλλά δεν έχουν προχωρήσει αρκετά σε άλλους τομείς. Αυτό λοιπόν το ενδιάμεσο βήμα και το γεγονός ότι τα σχέδια αυτά είναι προσχέδια μας έχει επιτρέψει να υποβάλουμε συγκεκριμένες συστάσεις και γι' αυτό είναι σημαντικές είναι σημαντικά τα σχέδια έκθεση, είναι όμως απλά σχέδια έκθεση. Πιο σημαντικό είναι το τι θα συμπεριλαμβάνεται τελικά στις εκθέσει. Είπαμε ότι τα εθνικά σχέδια είναι πολιτική δέσμευση, είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω να εξετάσουμε και την νομοθεσία που υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία. Έχουμε λοιπόν μια σειρά εργαλείων, όπω έχουμε πάντα στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, για να διασφαλίσουμε την σωστή εφαρμογή και να φροντίσουμε τα κράτη-μέλη να πληρώσουν τι υποχρεώσει που έχουν αναλάβει ω μέρο αυτή τη διαδικασία αυτή. Μεσοπρόθεσμα το πιο σημαντικό είναι η στενή επαφή με τα κράτη-μέλη για να πετύχουμε τις βελτιώσεις που ζητήσαμε και να δούμε ε, να εντείνονται οι προσπάθειες όσον αφορά τα εθνικά σχέδια και σε τεχνικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο και ε, στο Συμβούλιο Ενέργειας ε, αυτό το μήνα γίνονται πολλές προσπάθειες και γίνεται πολλή δουλειά. Θα πρέπει να δούμε οι τελικές εκθέσεις που θα μα φτάσουν, πού βρισκόμαστε όσον αφορά την επιτεύξη των στόχων, πού βρισκόμαστε όσον αφορά το επίπεδο φιλοδοξία, πού βρισκόμαστε όσον αφορά συγκεκριμένα ε, μέτρα και ε, ε, προγράμματα και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τελικά την κατάσταση. Επανέρχομαι στους πολίτες. Κάποιοι από εσά αναφέρθηκαν ε, στην ενεργειακή ένδια που παραμένει σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Υπάρχουν διάφορες ανησυχίες σε διάφορα κράτη-μέλη και σε διάφορα κράτη-μέλη και σε διάφορες περιφέρειες τους. Είδαμε λοιπόν ε, κάποιες αντιδράσεις σε κάποιες από τις πρωτοβουλίες. Υπήρξαν ανησυχίες σχετικά με τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο κάποιων ε, πρωτοβουλειών. Στις πολιτικές κατευθυντήρες γραμμές αναφέρεται μία δίκαιη μετάβαση, τον αλλημάνων υπόψη διάφορες κοινωνικές ομάδες. Έτσι λοιπόν έχουμε όλοι μία σαφή κατεύθυνση, έναν σαφή προσανατολισμό και όπως είπα προσλέπω στη συνεργασία μαζί σας πάνω στα θέματα αυτά. Τέθηκε ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή και εάν η νέα πράσινη συμφωνία και το όραμα που περιγράφεται ε, στις πολιτικές κατευθυντήρε γραμμές έχει μόνο να κάνει με την εφαρμογή ε, της υιοθετημένης ε, νομοθεσίας ή το αν θα υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες, νομίζω ότι είναι σαφέ στι πολιτικέ κατευθύνσει γραμμέ ότι θα περιμένουμε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε, ένα νόμο για το κλίμα, ένα ταμείο για τη δίκαιη μετάβαση. Θα υπάρξουν λοιπόν νέε πρωτοβουλίες. Σε οτιδήποτε κάνουμε θα πρέπει να βασιζόμαστε στην σωστή εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. τέθηκε ερώτηση σχετικά με το τέλος ε, για τον άνθρακα και δεν ξέχασα να απαντήσω πριν. Έχω περάσει πολύ καιρό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σκεπτόμενη, προβληματιζόμενη πάνω στο θέμα αυτό. Τα επόμενα χρόνια θα ασχοληθώ ακόμα περισσότερο με το θέμα, διότι... Πράγματι είναι ένα θέμα που θίγεται στις πολιτικές κατευθυντήρες γραμμές. Δεν μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένη σχετικά με το πού και πότε διότι θα απαιτήσει προσεκτική ανάλυση και καλή προετοιμασία από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να αναλυθούν οι διάφορες πτυχές και όσον αφορά την ε, μετεγκατάσταση των εκπομπών, θα πρέπει να εξεταστούν όμως και οι οικονομικές συνέπειες ε, καθώς και εθνικά ζητήματα όσον αφορά με τις διεθνείς δεσμεύσεις μας. Ε, θα υπάρξει λοιπόν κάτι συγκεκριμένο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να, σας, να είμαι πιο σαφής να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με την αποθήκευση, την καινοτομία, την τεχνολογία και σχετικά με την σύζευση των διαφορών τομέων. Ε, τι θα κάνουμε ε, για να το πετύχουμε αυτό. Νομίζω ότι βρισκόμαστε ακόμη σε ένα αρχικό στάδιο χαρτογράφησης αυτή η ολοκλήρωση των διαφορών τομέων, η σύζευση των διαφορών τομέων ε, έχει διαφορετική σημασία για διάφορους ανθρώπους. Θα πρέπει να χαρτογραφήσουμε τα διάφορα στοιχεία που χρειαζόμαστε και νομίζω ότι λίγα λέω όταν λέω ότι είναι πολύπλοκο το θέμα. Πρέπει να εξετάσουμε τις διάφορες πηγές ενέργειας. Είναι εξορισμού δύσκολο το θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε προσεκτικά. Υπάρχει επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο τεχνολογίας, αποθήκευση, υδρογόνο. Η τεχνολογία λοιπόν είναι η μία πλευρά της λύσης, αλλά και η ένταξη των τεχνολογιών στη βιομηχανία μας, στην οικονομία μας, ε, για να είμαστε και ανταγωνιστικοί, ε, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό, προσβλέπω στην επόμενη συζήτηση μαζί σας. Επίσης, ε, τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και ιδιαίτερα για την ε, στέγαση, για τις κατοικίες. Ε, η ενεργειακή απόδοση εμπεριέχει ε, απίστευτες δυνατότητες, αλλά είναι απογοητευτικό το πόσο λίγη πρόοδο έχουμε σημειώσει στο θέμα αυτό. Αν εξετάσετε τα κτίρια στην Ευρώπη, θα διαπιστώσετε ότι ε, είμαστε μία ήπειρος με πολύ όμορφα παλαιά κτίρια. Θα πρέπει όμως να δούμε πώς μπορούμε να τα κάνουμε πιο ενεργειακά αποδοτικά. Χρειάζονται λοιπόν επενδύσεις. και θα χρειαστεί και ε, δημόσια χρηματοδότηση αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και τη σχέση ανάμεσα στους διάφορους τομείς πολιτικής, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Και νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα από τα σημερινά θέματα. Ε, όπως σας είπα όμως, ε, σε όσα δεν απάντησα σήμερα, πολύ ευχαρίστω ε, θα απαντήσω στο μέλλον. Α, όχι, όχι, τελευταία, τελευταία παρατήρηση. Τέθηκαν συγκεκριμένες ερωτήσεις, ε, συγκεκριμένα ε, εθνικά θέματα, την ΔΕΗ στην Ελλάδα, ε, την υπόθεση Χάντρο στη Γαλλία και τις επιδοτήσεις ε, για ορυκτά καύσιμα σε κάποια κράτη-μέλη. Κάποιες υποθέσεις τις γνωρίζω από την προηγούμενη μου θέση, αλλά δεν νομίζω ότι ενδείχνεται να συζητήσω αυτά που γνωρίζω από την προηγούμενη μου θέση εδώ. Είναι όμως συγκεκριμένα εθνικά θέματα τα οποία όπως σας είπα τα γνωρίζω από την προηγούμενη μου ε, δουλειά, αλλά συνεχίζω να ασχολούμαι με αυτά εξετάζοντας τα υπό το των διαφόρων στόχων μας, ε, την ενεργειακή ασφάλεια, τους ε, στόχους μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λοιπά. Όσον αφορά το θέμα των ορυκτών καυσίμων, όπως σας είπα, είναι κάτι που εμπεριέχεται στα εθνικά ενεργειακά και κλιματικά σχέδια. Σε όσα κράτη-μέλη δεν μας έχουν πει τι στοχεύουν να κάνουν όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα, έχουμε επανέλθει και έχουμε ζητήσει να είναι πιο συγκεκριμένα. Θα κλείσω εδώ, διότι είναι πολύ περασμένη ώρα. Σας ευχαριστώ όμως πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε και για μια πολύ καλή πρώτη συζήτηση. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ, σας ευχαριστώ συνάδελφοι για το ενδιαφέρον σας και χρειαζόμαστε μια πολύ αποτελεσματική Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Ε, έχουμε πολλές ελπίδες ε, και ελπίζουμε να ξανασυναντηθούμε όσο γίνεται το σύντομότερο για να συζητήσουμε τα άλλα ζητήματα. Συνάδελφοι, δεν έχει λήξει ακόμα η συνεδρίαση. Εδώ και ώρες ακούω τα όσα λέτε. Δέκα δευτερόλεπτα λοιπόν δώστε μου για να κλείσω τη συνεδρίαση. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί 25-26 Σεπτεμβρίου. Λήξη τη σημερινή συνεδρία. Σας ευχαριστώ θερμά.